Bonjour à tous, merci de prendre place. Καθίστε παρακαλώ, είναι 9 και 5. Έφτασε η στιγμή να ξεκινήσουμε. Η σωστή συνεδρίαση είναι αυτή που ξεκινά στην ώρα της. Πάντα το λέμε αυτό. Ε, voilà. Λοιπόν. Vous plaît, je λοιπόν, σας παρακαλώ, καθίστε γιατί πρόκειται να ξεκινήσουμε. Ο, γενικό ο Γενικός Διευθυντής θα έρθει, όμως η ώρα είναι 9 και 5 και αρχίζουμε στις 9. Αν τρώμε το χρόνο μας και δεν σταματήσουμε εγκαίρως ε, θα παραπονιέστε. Λοιπόν, ξεκινάμε για αποσεβασμό και μόνο σε αυτούς που έχουν έρθει στην ώρα τους. Οπότε έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε τον κύριο Φωτιά στην Επιτροπή μας, ο οποίος αν δεν είναι εδώ θα έρθει σε λίγο, είναι Γενικής Διεύθυνσης ε, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΦΚΟ, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προέκυψε από την συγχώνευση της Γενικής διεύθυνση ΔΕΒ και της ΑΙΚΟ. Ο κύριος ε, Φωτιάδης έγινε τον Ιούλιο του 2010 ε, Γενικός Διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης μετά από μακρά πορεία στην Κομισιόν όπου ήταν Γενικός Διευθυντής για τις αλλάσεις υποθέσεις στην Αλία και προηγουμένως βοηθός Γενικού Διευθυντή για τις εξωτερικές σχέσεις. Ο βασικός λόγος για τον οποίο χρειάστηκε να περιμένουμε ένα χρόνο περίπου μετά την, το διορισμό του για να έχουμε τη χαρά να τον συναντήσουμε εδώ είναι ότι στο διάστημα αυτό έγιναν σημαντικές αλλαγές στην δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με τη δημιουργία της SUAE, ένα μέρος του ε, προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης DEV και της ICO ε, ε, δημιούργησαν τη νέα Γενική Διεύθυνση DEVCO, η οποία είναι πλέον απαραίτητο να να αναδιοργανώσει και να διαμορφώσει το έργο της. Ο κύριος Φωτιάδης έχει φτάσει. Φτάνει, έρχεται. Θα του δώσουμε το λόγο όταν έρθει στην αίθουσα. Οπότε... κάνω μία μικρή ε, διόρθωση στον κατάλογο ψηφοφοριών που έχετε ε, για την παράγραφο 8 η τροπολογία 67 θα καταπέσει αν εγκριθεί η 68. Αυτό εγκρίθηκε με την τροπολογία 65. Επαναλαμβάνω. Μικρή διόρθωση. Στην παράγραφο 8. Η 67 θα καταπέσει αν η 66 εγκριθεί και όχι η 65, η 66. Οπότε θα δώσουμε πλέον το λόγο, ε, θα τον αφήσω να πιει και λίγο νερό, στον κύριο Φωτιάδη τον οποίο ε, προλίγου σας ε, παρουσίασα. Κύριε Φωτιάδη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Έχει περάσει ένα διάστημα από την εποχή που διορίστηκα στην πρώην ΔΕΒ, εδώ και ένα χρόνο περίπου. Το διάστημα, στο διάστημα αυτό συνέβησαν πολλά και γι' αυτά θα ήθελα να σας μιλήσω. Έχω δίπλα μου τον Λουκ Μπαμπύρ, ο οποίος με βοήθησε να στήσω τη νέα αυτή οργανωτική δομή. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν εν συντομία την τη γενική αυτή διεύθυνση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ξέχασα τα γυαλιά μου. Σε παρακαλώ Λουκ μπορείς να παρουσιάσεις το οργανόγραμμα διότι δεν μπορώ να το διαβάσω, ζητώ συγγνώμη. Και επειδή επειδή είναι αυτή η οργανωτική δομή προέκυψε ε, ε, να έχει 1.400 άτομα και 3.000 άτομα σε αντιπροσωπείες ε, είναι αρκετά ε, ογκώδης, είναι σοκ να το βλέπει κανείς αυτό μπροστά του. Αποτελείται περίπου από 50 μονάδες. Θα σας διανύμω λοιπόν το οργανόγραμμα για να το διατρέξουμε μαζί. Θα σας κάνω μία παρουσίαση, στην οποία όμως φοβάμαι όπου δεν, ότι δεν θα μπορείτε να διαβάζετε τους τίτλους. Οπότε ας δούμε από κοινού το οργανόγραμμα και κατόπιν ας επιστρέψουμε ε, στους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή η συγχώνευση, τι κάναμε και ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτύχει αυτή η Γενική Διεύθυνση. Σας παρακαλώ να προβάλλετε το οργανόγραμμα. Δεν μπορεί να προβληθεί. Εντάξει. Λοιπόν, πάρτε τον μπροστά σας και θα το διατρέξουμε. Το κόκκινο είναι αυτό το οποίο γνωρίζετε και από παλιά. ΑΕΤΚΟ, η δημιουργία της ε, ΑΕΤΚΟ. Είναι οι τέσσερις περιφερειακές διευθύνσεις που έχουν την ευθύνη της υλοποίησης της βοήθειας και επίσης αναλαμβάνουν την οικονομική ευθύνη της διαχείρισης ε, των πόρων για τα προγράμματα. Είναι δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια συνολική εικόνα του πώς ε, διαχειρίζονται τα χρήματα οι 110 αντιπροσωπείες και πώς εφαρμόζουν τα προγράμματα. Έχουμε τέσσερις γεωγραφικές διευθύνσεις, η Ποσαχαρική Αφρική και ε, οριζόντια ζητήματα ΑΚΕ. Μετά υπάρχει η πολιτική γειτονίας, Βόρεια Αφρική και Ανατολική Ευρώπη, Κάφκασος. Λατινική Αμερική, Καραϊβική και Ασία, Κεντρική Ασία και Ειρηνικό. Ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά αυτής της γεωγραφική δομή, Ότι ουσιαστικά διαιρέσαμε την γεωγραφική διεύθυνση ΑΚΕ, δηλαδή η Καραϊβική εντάχθηκε με τη Λατινική Αμερική, Αμερική και ο Ειρηνικό έχει πάει στην Ασία. Για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί θέλαμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην υποσαχαρική Αφρική και θέλαμε να υπάρχει μια διεύθυνση που αποκλειστικά ασχολείται με την υποσαχαρική Αφρική λόγω της σημασίας της ε, με στην ανάπτυξη και προσθέσαμε την Καραϊβική στην ε, Λατινική Αμερική και τον Ειρηνικό στην Ασία γιατί θεωρήσαμε ότι από πολιτική, οικονομική και περιφερειακή σκοπιά τα οικονομικά και πολιτικά ζητήματα των χωρών αυτών εξαρτώνται περισσότερο από την περιοχή τους, από τη γειτονιά τους. Η Καραϊβική δηλαδή βρίσκεται υπό την ε, ισχυρή επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Λατινικής Αμερικής και αντίστοιχα ο Ειρηνικός από την Νότια Ανατολική Ασία. Αυτή είναι λοιπόν η δομή οποία, ε, με την οποία διανέμονται τα προγράμματα. Τώρα, σε αυτές τις τέσσερις διευθύνσεις υπάρχουν αυτά τα που σημειώνονται με κίτρινο ή με καφέ ολέ, όπως λέει ο μιλητής, είναι τα τμήματα των αντιπροσωπιών που συνδέονται με κάθε γεωγραφική διεύθυνση. Όπως σας είπα, όλοι όσοι εργάζονται στις αντιπροσωπείες ασχολούνται με την χρήση των κονδυλίων, περίπου 3.000 άτομα. Και τέλος, επιτέλους μετά από τόσα χρόνια, καταφέραμε αυτοί οι οποίοι να έχουν την ευθύνη της πολιτικής και την εφαρμογή της πολιτικής να είναι υπεύθυνοι και για την διαχείριση αυτών των αντιπροσωπιών που εκτελούν τα προγράμματα. Θα επανέλθω σε αυτό, είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Τώρα, τι άλλο ε, καινούργιο στοιχείο έχει αυτό το οργανόγραμμα. Αν κοιτάξετε το γαλάζιο κομμάτι, θα δείτε ότι υπάρχουν δύο διευθύνσεις ε, που είναι θεματικές. Η μία ασχολείται με την ανάπτυξη και την οικονομική ανάπτυξη και η άλλη που ασχολείται με την ανθρώπινη ανάπτυξη και την κοινωνική ανάπτυξη. Εκεί θα βρείτε όλους τους τομείς και τα διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και στα οποία θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Φερρυπίν η ανάπτυξη, η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάπτυξης έχει την αγροτική ανάπτυξη, πιστιστική ασφάλεια, περιβάλλον, τα χρηματοοικονομικά ε, μέσα είναι τα νέα μέσα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να εμπλακούν και οι ιδιώτες επενδυτές στην ανάπτυξη, ανάπτυξη ιδιωτικού τομέα, εμπόριο, ενέργεια και υποδομές όλα αυτά έχουν σχέση με την ανάπτυξη και την οικονομική ανάπτυξη και θα είναι στο προσκήνιο, θα είναι προτεραιότητες στη νέα δουλειά μας στο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργία θέσεων εργασία. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι, τα θέματα που είναι περισσότερο παραδοσιακά ανθρώπινης κοινωνίας, δημοκρατία, κοινωνία των πολιτών, απασχόληση, παιδεία και μια σειρά από άλλα. Κατόπιν υπάρχει μια διεύθυνση, η διεύθυνση Α, που θα ασχοληθεί με την αναπτυξιακή πολιτική. Δηλαδή η μονάδα διατύπωσης, διαμόρφωσης της πολιτικής, η οποία ασχολείται με την μελλοντική αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Πράσινη Βίβλο. Υπάρχει μια μονάδα που θα ασχοληθεί με την οικονομική ανάλυση, τα δημόσια οικονομικά και την ε, στήριξη, τη δημοσιονομική στήριξη. Είναι αυτοί που θα ολοκληρώσουν την ανακοίνωση τα περί του προϋπολογισμού. Υπάρχουν επίσης οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φροντίζουν οι συνάδελφοι στις άλλες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προωθήσουν τα θέματα αυτά, όλες οι τομεακές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή εμπόριο, μετανάστευση, ενέργεια, περιβάλλον κλπ να φροντίζουν στο μέλλον να συνεργάζονται με έναν τρόπο ώστε το τελικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα να είναι θετικό. Αυτά θέλει να κάνει λοιπόν η Γενική μας Διεύθυνση περαιτέρω. Θα υπάρξει μια νέα μονάδα, ένα νέο τμήμα το οποίο θα έχει σε στόχο την ανάπτυξη μιας ε, πρέπουσας πολιτικής για τις εύθραυστες χώρες και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κρίσεων. Εν τέλει, <clears throat> θα θέλαμε να δοθέσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα, στον αντίκτυπο των ενεργειών μας και στην διαφάνεια, όπως έχουμε υποσχεθεί πολλές φορές στο παρελθόν και θα είναι ένας από τους κύριους στόχους του, της Πρασίνης Βίβλου και γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει μια νέα διεύθυνση η οποία θα αντιμετωπίσει τα θέματα της πολιτικής μας και του αντικτύπου. Τέλος έχουμε και το, την διεύθυνση πόρων ανθρωπίνων τέ και αψύχων που βλέπετε στο δεξιό τμήμα είναι ο προπολογισμό, τα νομικά θέματα, λογιστικό έλεγχο, αλλά κυρίως και πρωτίστως η διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού. Έχουμε περίπου 1.500 άτομα στις Βρυξέλλε και 3.000 οι οποίοι εργάζονται σε αναπτυξιακά θέματα σε 110 αντιπροσωπείε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οργανόγραμμα λοιπόν αυτό σας δείχνει ότι υπάρχουν δύο αναπληρωτές γενικοί διευθυντές οι οποίοι θα βοηθούν την εργασία συντονισμού και θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη συνέχεια και συνοχή μεταξύ θεματικών, εθνικών και γεωγραφικών προγραμμάτων μέσα στην περιφερειακή μας αντιμετώπιση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία του νέου οργανογράμματος. και θα υπάρξουν και κάποιες ε, μονάδες, κάποια τμήματα τα οποία θα με αρρωγήσουν για να μπορέσω να έχω καλύτερο συντονισμό η μονάδα εσωτερικού λογιστικού ελέγχου κτλ. Λίγο πολύ έτσι διαγράφεται το σχήμα από την 1η Ιουνίου και επέκεινα. Λίγο φοβιστερό μπορεί να σας φαίνεται, αλλά νομίζω ότι έχουμε κάνει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια σαφήνεια σε σχέση με τους στόχους μας, σε σχέση με τις προτεραιότητές μας στο μέλλον για την ανάπτυξη πολιτικών και για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να τις φέρουμε σε πέρας. Έχουν διεξέλθει αυτό το έγγραφο, θα ήθελα τώρα να σας εξηγήσω γιατί κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες. Καταρχήν, ο στόχος μας ήταν να συνενώσουμε και πάλι τον σχεδιασμό της πολιτικής και την εφαρμογή της, και να μην υπάρχει τεχνητή ε, διάκριση όπως ήταν μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΒ και της Γενικής Διεύθυνσης ΑΙΤΚΟ, μια τεχνητή διαίρεση η οποία διήρκησε πολλά χρόνια ΦΕΦ. Είναι καιρό επιτέλους να έλθουν μαζί και να συνεργαστούν αυτές οι δύο <clears throat> γενικές διευθύνσεις γιατί πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι αναπτύσσουν τις πολιτικές θα πρέπει να το κάνουν αναγνωρίζοντας τις πραγματικότητες και αναγνωρίζοντας την εμπειρία που έχει κτηθεί στην εφαρμογή των προγραμμάτων μας, αλλιώς κανείς δεν πρόκειται να λάβει υπόψη αυτά τα οποία πράττομεν και τούμπαλιν. Και επίσης αυτοί οι οποίοι εφαρμόζουν τα προγράμματα θα πρέπει να γνωρίσουν ποια είναι τα πολιτικά ε, ζητούμενα και διακυβευόμενα, ποιοι είναι οι στόχοι που επιζητούμε μέσα από τα σχέδια και τα προγράμματά μας. Κατά δεύτερο λόγο, θέλουμε να συγκεντρώσουμε τις δεξιότητες σε μια γενική διεύθυνση για να δημιουργήσουμε ένα κέντρο αριστείας και στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή των πολιτικών συνεργασίας και ανάπτυξης. Τρίτον, ποιον θα παίρνουν στο τηλέφωνο οι άνθρωποι όταν θέλουν να μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Αυτό ήταν πολύ μπερδεμένο. στο παρελθόν υπήρχαν πάρα πολλές ε, Υπηρεσίε δύο διαφορετικέ γενικέ διευθύνσει. Ήταν διαφορετικά τα μηνύματα που δίνανε για το ίδιο θέμα. Γι' αυτό θέλαμε να έχουμε ένα μονάχα σημείο εισόδου για όλες τις ερωτήσεις που αφορούν την ανάπτυξη και ένα μονάχα σημείο αναφοράς για τον έξω κόσμο. Αν μπορώ τώρα να πάω στο δεύτερο, στη δεύτερη διαφάνεια για τα θέματα αυτά, ήταν πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι <clears throat> υπάρχουν κοινά μηνύματα τα οποία δίδουν όλες οι αντιπροσωπείες μας, να υπάρχει σωστή επικοινωνία. Φανταστείτε να θέλει κάποιος να πάρει μια απόφαση και να πρέπει να έρθει σε επαφή και να συμβουλευτεί δύο γενικούς διευθυντές χωρίς καμία εγγύηση ότι το μήνυμα που θα πάρουν από τις δύο γενικές διευθύνσεις θα ήταν συνεκτικό. Θέλαμε επίση να έχουμε μονάχα ένα συνομιλητή για την εξωτερική υπηρεσία <coughs> και εναντί της Κομισιόν, ώστε να υπάρξει συνοχή και συνέχεια για την εξωτερική δράση και συγχρόνως να υπάρξει πολιτική συνεκτικότητα στην ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταίο αλλά όχι ίστατο και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, θέλαμε να ξεπεράσουμε την επικάλυψη σε επίπεδο προσωπικού για να απελευθερώσουμε ένα αριθμό υπαλλήλων οι οποίοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις και τις δυσκολίες που είχαμε στο σχεδιασμό της πολιτικής αλλά και στην εφαρμογή της και να τους επιτρέψουμε να αντιμετωπίσουν τις νέες εγυρώμενες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η γενική μας διεύθυνση. Ποιε αυτέ είναι προκλήσεις όμως. Δεν πρόκειται εδώ να αναφέρω τις υπάρχουσες προκλήσεις, μόνο τις μελλοντικές. Τι πρέπει να κάνει η Γενική μας Διεύθυνση. Πρέπει να αναπτύξουμε ένα γενικό σχέδιο, μια πολιτική ανάπτυξη η οποία θα αφορά όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο και όχι μόνο την Αφρική. Και μια γενική τομεακή πολιτική ανάπτυξης για τους τομείς που έχουν μεγάλη επίπτωση στα θέματα ανάπτυξης. Δεύτερον, θέλαμε να σχεδιάσουμε μελλοντικές πολιτικές ανανεώνοντας, εξυγχρονίζοντας τις πολιτικές μας ανάπτυξης ε, και φυσικά να έχουμε τα στοιχεία τα οποία θα εισρεύσουν στην πολιετή δημοσιονομική σχεδίαση σημείο 4 του προπολογισμού. Παραδείγματος χάρη. Τρίτον, θα πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι η ευρωπαϊκή εν γέννη διάσταση, εξασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη είναι τμήμα μιας συνεκτικής εξωτερικής δράσης. δύο συνεργαζόμενοι, όταν συνεργαζόμαστε με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, να εξασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές κατατομής είναι τμήμα μιας συνεκτικής πολιτικής ανάπτυξης, και τέλος θέλουμε να δώσουμε μια συμβολή στην αντιμετώπιση των παγκοσμίων προκλήσεων κτλ. Και φυσικά να παίξουμε ρόλο στην ε, υποστήριξη στόχων σε παγκόσμιο επίπεδο και την παγκόσμια διπλωματία για την ανάπτυξη και το συντονισμό με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης για μια συνεκτική εξωτερική πολιτική. 3.000 υπαλλήλους έχουμε σε 110 αντιπροσωπείες ανά τον κόσμο και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις ευθύνες μας έναντι αυτών των ατόμων. Αυτό είναι σημαντικός πρόσθετος φόρτος εργασίας. Τελευταίο σημείο το οποίο θέλω να σας αναφέρω. Έχουμε πλέον τα μέσα και την διοικητική εξουσία για να εξασφαλίσουμε κάτι το οποίο έχει καθυστερήσει πολλά χρόνια, την επανεξισορρόψη του αριθμού των ατόμων στις διάφορες αντιπροσωπείες. Ξέρετε ότι η κατανομή αυτή στις διάφορες αντιπροσωπείες είναι αποτέλεσμα του ρού της ιστορίας. Είναι μια συσσόρευση ιστορικών γεγονότων που δεν είχαν πάντα να κάνουν με την αποτελεσματικότητα. Τώρα θέλουμε να επανεξετάσουμε το φόρτο εργασίας των αντιπροσωπιών για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε την επαρκή στελέχωση εκεί που είναι απαραίτητη, αριθμητικά και σε επίπεδο δεξιοτήτων, αλλά και προφιλικά το οποίο σημαίνει αυτή τη στιγμή και πρέπει να εξασφαλίσουμε περαιτέρω ότι θα έχουμε άτομα και πόρους που θα μπορούν να είναι εκεί όπου είναι πλέον πρόσφοροι και χρήσιμοι και όχι να είναι εκεί που δεν τους χρειαζόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας ε, παρουσιάσω υπομορφή εισαγωγή και φυσικά εδώ είμαι και θα απαντήσω και τα ερωτήματά σας. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να λάβει χώρα αυτό το εγχείρημα με τις λιγότερες δυνατέ διαταραχές και τριβές σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των αρμοδίων γενικών διευθύνσεων, γιατί φυσικά προέχει να μπορεί να γίνεται με σωστό τρόπο η εκτέλεση του προϋπολογισμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων να συνεχίζουν απρόσκοπτα και αμέριμνα. <clears throat> Διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα νέο πλαίσιο δημοσιονομικών προοπτικών και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η αποτελεσματικότητα της γενικής μας διευθύνσεως δεν θα τεθεί εν αμφιβόλο και απλώς σας υπενθυμίζω ότι αν στο τέλος του έτους δεν είμαστε σε θέση να καταδείξουμε θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις υποχρεώσεων και πληρωμών, θα τη βρουν οι αρχηγοί των οικονομικών, οι Υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών και θα θεωρήσουν ότι δεν είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στους ε, δημοσιονομικούς στόχους της Κομισιόν. Και υπάρχει πραγματικά η αίτηση από εμάς να έχουμε περισσότερα χρήματα για την ανάπτυξη. Αν δεν το καταδείξουμε αυτό ότι είναι απαραίτητα περισσότερα χρήματα με μια σωστή εκτέλεση του προπολογισμού, τότε θα χάσουμε το παιχνίδι. Προσπαθούμε λοιπόν να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα με τρόπο που θα οδηγήσει σε στις λιγότερες νατές αναταράξεις, αλλά ένα εγχείρημα αυτού του μεγέθους δεν μπορεί να γίνει ποτέ χωρίς να υπάρξουν κάποια άτομα τα οποία θα δυσφορήσουν και θα δυστροπήσουν ακόμα και αν η πλειοψηφία αναγνωρίζει τη σημασία και την χρησιμότητα του εγχειρήματο. Προσπαθούμε λοιπόν να το κάνουμε με ένα τέτοιο τρόπο που θα λάβει υπόψη τις επιθυμίες όλων των συναδέλφων, ακόμα και αυτών οι οποίοι δεν θα είναι απόλυτα ικανοποιημένοι. Εμείς ακούσαμε την άποψη πολλών συναδέλφων, προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη τις επιθυμίες τους κτλ. Αυτά λοιπόν. 1η Ιουνίου ξεκινάει το νέο σχήμα και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να κάνουμε τα πράγματα, πολύ καλύτερος σε σχέση με το παρελθόν και είναι η ειλικρινής μου ελπίς ότι το εγχείρημα θα στεφθεί υπό επιτυχίας και έτσι θα υποστηρίξουμε πλήρως τη στρατηγική που διέρχεται το νέο αυτό οργανόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στους, ε, στα σχόλια των μελών της Επιτροπής. Ο κύριος Γκέρεν, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας έκανε την παρουσίαση αυτή. Τόσο πρωί κιόλα, ακόμη δεν έχει. έχει. Έχει ανοίξει το μυαλό μας πρωί-πρωί, είμαστε φρέσκοι και μπορούμε να καταλάβουμε όλες τις αποχρώσεις του μήνυματός τους. Νομίζω ότι μάλιστα κατάλαβα ορισμένα μηνύματα τα οποία δημιουργούν και ερωτήματα από πλευρά. μου. Σε ποιο βαθμό το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η διάκριση μεταξύ των ΑΚΕ ε, είχε κάποιο νόημα σε σχέση με την προετοιμασία αυτής της διαδικασίας γιατί είναι γεγονός ότι οι ΑΚΕ συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μιας σύμβασης. Τώρα, το να γίνει μια κατηγοριοποίηση των χωρών και σε τρία διαφορετικά τμήματα, ε, μήπως αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα συνοχής και συνέπεια στην προσέγγιση μας προς τις χώρες αυτές, γιατί δεν είναι τα ίδια άτομα που ασχολούνται με το ίδιο φάκελο. Ε, ενώ τα συμφέροντα ε, των χωρών αυτών ε, είναι τέτοια που καλό θα ήταν να τις μεταχειριζόμαστε με ομοιόμορφο τρόπο. Ενδεχομένως να είμαι και ένας από τους μόνους που ε, θέτουν αυτό το ερώτημα. γιατί την ιδέα αυτή την πήρε από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίοι στην αρχή της ε, συγχώνευσης ε, της ε, DGDEV με την DGEDCO είχαν προτείνει έναν προβληματισμό, ένα κέντρο προβληματισμού, τεκμηρίωσης και προτάσεων ανεξάρτητο. Ένα ανεξάρτητο κέντρο και νομίζω ότι αυτό πραγματικά λείπει μου κάνει εντύπωση, για, μου κάνει ε, ο αριθμός των ατόμων που καταφέρατε να ε, χωρέσετε στα διάφορα σημεία του οργανογράμματός σας. Ε, οι περισσότερες από τις ιδιότητες τους έχουν να κάνουν με την καθημερινή δουλειά μας, με το daily business. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ απαιτητική η κατάσταση. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει δίπλα ένα κέντρο το οποίο θα έχει χρόνο και θα μπορεί να αντιμετωπίζει αυτό το φόρτο της καθημερινής εργασίας, να προβληματίζεται για, τις στρατηγικές, ε, για τους στρατηγικούς προβληματισμούς. Ε. Και ένα ακόμη ερώτημα και τελευταίο που θα ήθελα να σας ε, θέσω. Η Lady Άστον, σε περίπτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων σύγκρουση μεταξύ των διαφόρων προπολογισμών, ε, μεταξύ ε, των, των διαφόρων προσανατολισμών, μεταξύ των υπευθύνων του οργανογράμματος αυτού, πώς θα, πώς θα γίνουν τα πράγματα. Γιατί, να σας πω ένα παράδειγμα που μπορεί να προκύψει στους επόμενους μήνες. Βλέπω εδώ, για παράδειγμα, την πολιτική που αφορά τις χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν να αντιμετωπίσουν εξέγερση του πληθυσμού. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Μπορεί να είναι θετικό το ότι κατηγοριοποιούνται όλα αυτά τα ζητήματα σε ένα συγκεκριμένο τμήμα ε, όσον αφορά, για παράδειγμα, ε, του κύκλου εργασίας. Ε, μήπως όμως υπάρχει και κάποιος κίνδυνος κατακαιρματισμού των πολύ συγκεκριμένων αναγκών που μέσω της αναπτυξιακής πολιτικής, πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας έχει κάποιο αποτέλεσμα για τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Ευχαριστώ. Θέλετε να ακούσουμε πολλές ερωτήσεις ή θέλετε να απαντήσετε σε αυτήν. Ο κύριος Πόγκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Διευθυντά, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Θα θέσω ένα θέμα που γνωρίζετε πολύ καλά, ε, την Task Force ε, PTOM στο πλαίσιο της DEFCO. Είναι ένα ζήτημα το οποίο άπτεται τη σημερινή σα παρουσίαση γιατί έχει να κάνει με το κομμάτι των χωρών ΑΚΕ, με αυτό το κομμάτι του οργανογράμματος. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω την εξή ερώτηση. Μου φαίνεται ότι αντιφάσκουν αυτά με τη νέα στρατηγική που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις ε, ΠΤΟΜ. Υπάρχει μια νέα εταιρική σχέση ε, που θα, συνδέ, θα αυξήσει τους δεσμούς με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο Επίτροπος Πίμπαλ στην τελευταία φορά στη διάσκεψη Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΤΟΜ ε, ανέφερε σε μια νέα εταιρική σχέση συνεργασίας όπως επίσης και για τη σημασία της σχέσης αυτής στο βαθμό που αυτά τα εδάφη είναι τμήματα της ευρωπαϊκής οικογένειας να ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Γνωρίζετε ότι βρίσκονται σε διάφορα ε, σημεία των ωκεανών, ε, ε, σε μια δύσκολη γεωγραφική θέση και νομίζω ότι δεν καλύπτονται με, τον, με το τρέχον οργανόγραμμα όλα αυτά τα εδάφη. Νομίζω λοιπόν ότι η Task Force ε, θα βρίσκεται σε μια θεματική ενότητα ε, στο πλαίσιο της, ε, όπως για παράδειγμα η ΡΟΥΠ στην Γενική Διεύθυνση Περιφερειών και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ενίσχυση του διαλόγου του διεθνούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci, Monsieur Ponga. Vous voulez déjà répondre Θέλετε να απαντήσετε? Ναι. Ευχαριστώ. Για το ερώτημα του κυρίου Γκέρενς. Ναι, υπάρχουν ε, μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα στο να είναι σε μία διεύθυνση η ΑΚΕ. Ένα ε, μειονέκτημα είναι βέβαια ότι οι ΑΚΕ, οι χώρες ΑΚΕ δεν έχουν υποχρεωτικά τις ίδιες ε, προτεραιότητες και, τις ίδιες, ε, και τους ίδιους στόχους. Δηλαδή άλλο η Ποσαχάρια Αφρική και ε, άλλο οι υπόλοιπε χώρες είναι χιλιάδες χιλιόμετρα η απόσταση παρά το γεγονός ότι είναι η κοινή πολιτική που έχουμε προς τις χώρες αυτές. Υπάρχουν λοιπόν υπέρ και κατά. Το συζητήσαμε με πρέσβη στον χωρών ΑΚΕ πολλές φορές και εξηγήσαμε ότι η το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η διάκριση και η διαφορετική κατηγοριοποίηση δεν σημαίνει ότι ε, θα έχουν χαμηλότερη προτεραιότητα σε σχέση με τα ζητήματα και διότι υπάρχουν και ορισμένα οριζόντια ζητήματα ε, που ασχολούνται για παράδειγμα και με την υποσαχάρη Αφρική και με τις υπόλοιπες χώρες ΑΚΕ ώστε να υπάρχει εξασφάλιση του συντονισμού σε σχέση με τα ζητήματα ΑΚΕ μεταξύ των ε, μεγάλων γεωγραφικών ε, ε, διευθύνσεων που θα έχουν την ευθύνη. Οπότε... Είναι ένας διαφορετικός τρόπος απλώς οργάνωσης. Έπρεπε να εξηγήσουμε στις χώρες ΑΚΕ ότι αυτό δεν σημαίνει επουδενή ότι δεν δίνουμε την ίδια σημασία όπως προηγουμένως στις χώρες ΑΚΕ. Όμως νομίζουμε από την άλλη ότι ήταν πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα ότι θα επικεντρωθούμε στην υποσαχάρια Αφρική με πιο αισθητό τρόπο. Και αυτό ήταν και ο λόγος ε, αυτής της αλλαγής. Όσον αφορά τώρα το κέντρο προβληματισμού που αναφέρατε, ναι, όντω το είχαμε σκεφτεί, αλλά σκεφτήκαμε ότι ίσω θα ήταν καλύτερα ο προβληματισμό αυτό να ενσωματωθεί στην, ε, στην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής ε, Πολιτικής. Πρόκειται γιατί για το τμήμα της διαμόρφωσης αναπτυξιακής πολιτικής. Ε, εκεί έγκυται Από το τμήμα αυτό περιμένουμε να μας δώσει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαμόρφωση της ε, ε, πολιτικής. Ε, το να έχουμε ένα κέντρο προβληματισμού ανεξάρτητο και εκτός των, του τμήματος αυτού δεν θεωρήσαμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο ο ανταγωνισμός τώρα μεταξύ των γειτονικών χωρών και των υπολείπων αναπτυσσομένων χωρών είναι γεγονός αυτό. Τι να κάνουμε, Εντάξει, δεν ήταν εύκολη απόφαση. Υπήρξε μια ε, μεγάλη συζήτηση ε, για το πώς θα αντιμετωπιστούν ε, τα ζητήματα στην Βόρεια Αφρική. Υπήρξε και μια ανακοίνωση με, για την Βόρεια Αφρική. Εχθές ο πρόεδρος μας είπε ότι δεν θα υπάρξουν κονδύλια που θα φερεθούν από χώρες που έχουν ε, ανάγκη τα κονδύλια αυτά. Όλα τα κονδύλια θα προκύψουν ε, από ε, τομείς που δεν χρειάζονται τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει από χώρες που δεν χρειάζονται πλέον κονδύλια αναπτυξιακή βοήθειας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ανακοινώσαμε και στην Πράσινη Βίβλο για την Ανάπτυξη. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει και ε, στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δημοσιονομικές προοπτικές και αυτό είναι κάτι που ε, αναφέρθηκε και χθε, όπως είπα, 1,2 δισεκατομμύρια επιπλέον για, τις, ε, για την πολιτική γειτονία είναι κάτι το οποίο πραγματικά σκοπό έχει να συμπληρώσει αυτή τη νέα προσέγγιση την οποία θέλουμε να έχουμε. Όσον αφορά το ζήτημα που έθεσε ο κύριος Πόγκα. Κοιτάξτε, εγώ περισσότερο χρόνο ε, περνάω στα μικρά υπερπόντια ε, διαμερίσματα, ε, οπότε τα γνωρίζω, ίσως περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Και πράγματι αναρωτιόμαστε αυτή τη στιγμή, προβληματιζόμαστε ποιο είναι το καλύτερο χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα υπερπόντια αυτά εδάφη Θα δούμε τι εναλλακτικέ ε, επιλογές έχουμε. Για μας το θέμα της Task Force δεν είναι ένα ε, μόνιμο ζήτημα. Οι νέες δημοσιονομικές ε, προοπτικές για τα υπερπόντια διαμερίσματα και εδάφη θα καθορίσουν ποια θα είναι αυτή η task force, κατά πόσο θα παραμείνει στην ε, δική μας ε, Γενική Διεύθυνση ή αν θα μεταφερθεί στη Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο ε, εξαρτάται από το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θα, θα επιζητήσουμε. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. 20 λεπτά μας μένουν. Το λέω για πρακτικούς λόγους γιατί έχω ακόμη 5 ομιλητές και θα ήθελα να είστε σύντομοι. Ο κύριος Φωτιάδης και αυτός θα πρέπει να μιλήσει συμπερασματικά και όσοι έχετε ξεχάσει την κάρτα της ψηφοφορίας σας να πάτε γρήγορα να την πάρετε γιατί θα σας χρειαστεί. Ο λόγο έχει ο κύριος Μπέργμαν. Ευχαριστώ πολύ. Μια παρατήρηση και μια ερώτηση. Παρατήρηση. Είναι εξαιρετικό το ότι όλες αυτές οι μονάδες που ασχολούνται με ανάπτυξη και συνεργασία έχουν συνδυαστεί κάτω από μια γενική διεύθυνση. Είναι πολύ καλό αυτό θα ενισχύσει τη θέση του Επιτρόπου Ανάπτυξης και ε, έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει και την πολιτική. Δεν είναι πάντως απαραίτητο να ε, δημιουργηθεί μια μονάδα μελέτης. Ε, αυτή η policy formulation του François Moreau είναι νομίζω πολύ καλή και εκεί γίνονται πράγματα σημαντικά, απαραίτητα. Τώρα η ερώτηση. Θέλω να, να ρωτήσω σε σχέση με αυτές τις μονάδες. Πώς ε, έχετε διαρθρώσει τις θεματικές μονάδες αφενός και τις ε, γεωγραφικές μονάδες ε, πώς συνεργάζονται, δηλαδή μπορεί κανείς να τα πει αυτά θεωρητικά αλλά στην πράξη πώς γίνεται. Και δεύτερον, Μπορείτε να μας δώσετε κάποια ιδέα για το, το τι θα εξοικονομήσετε πάνω κάτω με τη νέα αυτή οργανωτική δομή. Δηλαδή, για τα, από τα γενικά έξοδα, αυτά τα overhead costs που αφορούν την οργάνωση για παροχή αναπτυξιακής βοήθειας από την ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλες δύο και θα κλείσουμε. Κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Δεν έχω πιστεί απόλυτα ότι αυτή η αναδιανομή και η αναδιοργάνωση θα λειτουργήσει απρόσκοπτα. Κυρίως επειδή αυτό υποτίθεται ότι λειτουργεί από πρώτη έκτου και γι' αυτό δείξατε τον πίνακα άμεσα στην Επιτροπή. Παρά ταύτα, δεν νομίζω ότι είναι τόσο τελειωτική μορφή του και είμαστε ήδη τέλος Μαΐου. Έχω ερωτήσεις. Πόσες γυναίκες υπάρχουν ως βοηθοί γενικοί διευθυντές, ε, διευθύντριες και επικεφαλής τμήματων και δεύτερον, στην πράξη και στην λεπτομερός η συνεργασία μεταξύ της Υπηρεσίας Εξωτερικών, Εξωτερικής Δράσης και τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Πώς θα γίνει. Τέλος, Είπατε ότι πρόκειται να αφήσετε κάποιες χώρες. Ποιες θα είναι αυτές. Ευχαριστώ κυρία Κέλλερ, ο κύριος Ντεβά. Αν με συντομία παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Α, είναι μια ανάσα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ότι ήρθατε ε, ότι υπάρχει ένας ελέφαντας ε, στην αίθουσα και δεν το ονομάζουμε έτσι. Αν κάτι πρέπει να αλλάξει, ας αλλάξει. Επί πολλά χρόνια, δέκα χρόνια είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής και άκουγα ότι τα πάντα είναι θαύμα και τίποτα δεν χρειάζεται να αλλάξει, όλα πάνε πολύ καλά κλπ. Και, και, λοιπά. και τώρα έρχεται και μας λέτε ότι α, όχι, δεν πάνε καλά τα πράγματα, χρειάζεται αλλαγή. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά φυσικά δεν σταματώ εδώ. Αλλαγή ως προς τι Χθε ήρθε ο Άντρου Μίτσολ και μας είπε ότι αλλάζει τη DFID. Θα αρχίσει να κάνει πράγματα που δεν έχουν γίνει στο παρελθόν. Τα τελευταία 50 χρόνια, δεν ξέρω. Θα ξεκινήσει μετρώντας τις αποδόσεις και όχι το τι προσφέρεται. Είπε ότι θα εκπαιδεύσει 11 εκατομμύρια παιδιά φέτος με κόστος 20 ευρώ το κάθε παιδί και ότι πρόκειται να οικοδομήσει και να εφοδιάσει 19.000 νοσοκομεία ή ότι θα ανοίξει 10.000 πηγάδια. Δεν είπε, δεν θα λέω ότι θα ξοδέψω 600 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια. Θα έρχεται να μας λέει τι έχει κάνει, τι έχει αποδώσει. Έχουμε αλλάξει λοιπόν τους ανθρώπους, έχουμε αλλάξει το ρυθμό, το οργανόγραμμα. Το αποτέλεσμα θα αλλάξει. Η κυρία Τσίμερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πάντα όταν γίνεται μια αναδιάρθρωση σε επίπεδο οργανογράμματος αυτό σημαίνει είναι πρόδρομος ουσιαστικά μιας ουσιαστικής αναδιάρθρωσης σε σχέση με τους στόχους και τα εγχειρήματα. Και βλέπω ότι οι χώρες ΑΚΕ πηγαίνουν σε άλλες περιοχές γεωγραφικές ποια, ποιες θα είναι οι συνέπειες οι οποίες θα προκύψουν άμα δεν υπάρχουν όλες αυτές οι χώρες στο ίδιο τμήμα αλλά θα βρίσκονται σε διαφορετικές ε, σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ενώ είναι γεγονός ότι όλες καλύπτονται από την ίδια σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και, με τα ίδια, και συνδέονται με τα ίδια προγράμματα χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μήπως αυτό σημαίνει ότι εν καιρό θα υπάρξει μια αλλαγή και τη συνθήκη που διέπει τις σχέσεις μας με τις χώρες ΑΚΕ. Δηλαδή ότι η συνθήκη της ε, Σύμβαση Κοτονού θα αποτελέσει παρελθόν κάποια στιγμή δεύτερο ερώτημα το οποίο ήθελα να... Μάλλον πρωτού θέσω το ερώτημα. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό στην ε, τρίτη διεύθυνση σε της ΤΕΦΚΟ, ότι υπάρχουν και τέτοια σημεία τα οποία είναι στοιχεία θεματικά και ουσιαστικά. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να θέσω. Μας είπατε ότι βρίσκονται σε εναλλαγή. Εκ περιτροπή, αναλαμβάνουν την ε, διοίκηση των τμήματων ή επικεφαλής τμήματων. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Παρακαλώ, ό,τι θέλετε. Εντάξει, επιτρέψτε μου να... Πολλές ερωτήσεις, θα προσπαθήσω να απαντήσω στα γρήγορα γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Όσον αφορά τον το... το θέμα των αναπληρωτών, πρέπει να επανεξεταστεί η πρόσληψη των αναπληρωτών. Αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο περίπου, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν αναλάβει καθήκοντα. Είναι σημαντικό το ζήτημα γιατί αυτοί είναι αυτοί που πρέπει να εξασφαλίσουν το συντονισμό μεταξύ των θεματικών και των γεωγραφικών πολιτικών και προγραμμάτων. Τα γενικά έξοδα, αν έχουμε εξοικονομήσει χρήματα εκεί, σαφώς έχουμε επιστρέψει 50 θέσεις εργασίας προς την κεντρική υπηρεσία, τις οποίες η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει για άλλους λόγους. Και επιπλέον αυτή της οικονομία κλίμακας έχουμε εξοικονομήσει από το γεγονός ή μάλλον και ω εκ τούτου έχουμε κάνει οικονομίες που θα χρησιμοποιηθούν από άλλες θέσεις τη Γενική Διεύθυνση που θα κάνουν νέα πράγματα. Παραδείγματο χάρη, υπήρχαν γεωγραφικές διευθύνσει που αντιμετώπισαν σοβαρότατες δυσκολίες ε, πόρων. Έχουμε νέες θέσει ε, στην Αφρική, 20 νέε θέσει στην πολιτική γειτονία και πολλές θέσει για την διατύπωση πολιτική, τη, πολιτική στη διεύθυνση Α, όπως σας είπα, γιατί αρχικά σας είπα, η νέα γενική διεύθυνση πρέπει να αναπτύξει πολιτική για ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν κάνει σοβαρές οικονομίες κλίμακας και αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Τώρα, τα θεματικά προγράμματα. Πολύ καλή ερώτηση και καθόλου εύκολη. Μια ολόκληρη μέρα θα μπορούσα να μιλάω μόνο για αυτό το θέμα. Τα Οι θεματικές διευθύνσεις. Τι υποτίθεται ότι κάνουν. Τέσσερα πράγματα. Πρώτον, να αναπτύξουν πολιτικ... κλαδικές πολιτικές που να είναι πρωτοπόρες. Δεύτερον, να παρακολουθήσουν την εφαρμογή των διαφόρων κλαδικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιβάλλον και και να εξασφαλίσουν ότι θα είναι θετικό το αναπτυξιακό τους αποτέλεσμα. Δηλαδή στην εκτικότητα της πολιτικής τρίτων θα παρακολουθούν τις ε, αντιπροσωπείες και τις γεωγραφικές διευθύνσεις όσον αφορά τον προγραμματισμό τους. Και τέταρτον θα πρέπει να εκπονούν τα θεματικά προγράμματα που, στα οποία πηγαίνουν πολλά χρήματα. Θα κάνω αυτά τα τέσσερα πράγματα. Οπότε, ο συντονισμός με τις γεωγραφικές διευθύνσεις είναι απαραίτητος και απολύτως σημαντικός ανα πάσα στιγμή σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Αυτό ακόμα προσπαθούμε να το μελετήσουμε για να αποφασιστούν οι λεπτομέρειες της διαδικασίας που θα εφαρμοστεί. Και υπό την έννοια αυτή η Γενική Διεύθυνση είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την συνεργασία μεταξύ της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της ΤΕΒΚΟ. Πάλι και εδώ μια ολόκληρη μέρα δεν θα έφτανε για να σας τα πω όλα. Να το θέσω ως εξής. Πρέπει να πετύχουμε και να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή σχέση συνεργασίας με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβεί κάτι τέτοιο. Και πράγματι, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων σε επίπεδο γεωγραφικής μονάδας. Αυτές είναι εξαιρετικές γιατί και στο παρελθόν είχαν συνηθίσει να συνεργάζονται. Εκεί που ακόμα εκκρεμούν κάποια πράγματα είναι το θεσμικό επίπεδο. Ποιος δηλαδή θα αποφασίζει τελικά επί ποιου θέματος κλπ. Ξεκινώντας από τον προγραμματισμό και ε, προχωρώντας το τι, λέει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για την εφαρμογή προγραμμάτων και εάν αυτοί θα έχουν λόγο για το εάν και κατά πόσο θα πρέπει να γίνει μια πληρωμή για την στήριξη προπολογισμού μιας χώρας και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να ε, παίζουν και πολιτικά κριτήρια, να ε, το αν θα δαπανηθούν χρήματα για μια χώρα ή όχι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ποιο τελικά θα αποφασίζει για το ποιοι θα επανδρώνουν τι αντιπροσωπείε. Γιατί εγώ μεν έχω την διοικητική ευθύνη για αυτέ τι αντιπροσωπείε, όπω επίση και έχω την προσωπική ευθύνη για την σωστή διαχείριση των πόρων. Και οι άνθρωποι αυτοί ε, ε έχουν την ευθύνη να κάνουν αυτό το έργο εξ μου και τελικά στο τέλος του χρόνου μιλάμε, θα μιλάμε για 8 δισεκατομμύρια επιπλέον πόρους. Πώς λοιπόν θα μπορεί να μην έχω εγώ την, τον τελευταίο λόγο. Από την άλλη, εκείνοι έχουν την ευθύνη για την λειτουργία των αντιπροσωπιών. Πρέπει λοιπόν και αυτοί να έχουν ένα λόγο για το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, που πάνε κλπ. Αυτό είναι ένα θέμα που ακόμα πρέπει εκρεμεί. Θα λυθεί όμως. Εργανωτικά και λοιπά θέματα, ε, θεσμικά, είναι θέματα με τα οποία, για τα οποία συνεργαζόμαστε με την ε, υπηρεσία από την αρχή του χρόνου. Ο David Σάλιβαν και εγώ έχουμε κάνει μια σειρά από εβδομαδιαίες ε, συναντήσεις και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Τι ρώτησε ο κύριος Ντέβες. Α, ποιες χώρες θα, από, από ποιες χώρες θα φύγουμε. Δεν μπορώ τώρα να προκαταλάβω την ανακοίνωση της Κομισιόν, αλλά έχουμε διακηρύξει ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να δαπανούμε λίγα-λίγα τα χρήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμα και σε χώρες που οι ίδιες είναι δωρήτριες, ας πούμε η Κίνα, η Βραζιλία, χώρες που εντωμεταξύ έχουν ενταχθεί στην ομάδα των G20. Χώρες που έχουν αν, οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 10 ή του 20% ή που έχουν στρατιωτικές δαπάνες που είναι χιλιάδες φορές υψηλότερες από τα χρήματα που δίνουμε εμείς στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας. Οι χώρες που μπορούν να φροντίσουν τα αναπτυξιακά τους προβλήματα πολύ καλύτερα από ό,τι το, μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι χώρες αυτές μας έχουν πει ότι δεν ενδιαφέρονται για αυτή την αναπτυξιακή συνεργασία μαζί μας. Θέλουν να γίνεται μια συνεργασία σε ίση βάση επί ε, στρατηγικών κλαδικών θεμάτων κλπ. Εμείς ήμασταν αυτοί που επιμέναμε και αναγκάζαμε, τους αναγκάζαμε να δέχονται τα χρήματα που, που δίναμε. Επί πολλά χρόνια. Λοιπόν, θα αλλάξει αυτό. Αυτά τα χρήματα και οι πόροι, δηλαδή οι άνθρωποι που απασχολούνται στις αντιπροσωπείες για τις χώρες αυτές, θα φερεθούν από εκεί και θα πάνε κάπου αλλού σε χώρες που χρειάζονται περισσότερους ανθρώπους και περισσότερους πόρους να ασχοληθούν μαζί τους. Ο κύριος Ντέβα, ναι, θα κάνουμε μια αλλαγή επί τα βελτίο. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ότι πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να είμαστε σε θέση να επιδείξουμε σημαντικότερα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα όμως η Ένωση είναι υποχρεωμένη να έχει παρουσία παντού. Και αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να βρίσκεται και σε δύσκολες χώρες όπου το να δείξει κανείς ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι δύσκολο. Χώρες που η κατάσταση είναι λεπτή και που δεν μπορούμε να ε, ξεφύγουμε από κάποια όρια και εκεί είναι δύσκολο ε, να δείξουμε αποτελέσματα όπως δείχνουμε σε χώρες που λειτουργούν σωστά. Βεβαίω αυτή είναι η αρχή, αλλά η αρχή αυτή δεν εφαρμόζεται, δεν ισχύει για παντού. Γιατί αν ισχύει παντού θα διατρέχαμε έναν κίνδυνο να φύγουμε από τις δύσκολες χώρες. Διαφορετικοί κανονισμοί ε, για ΑΚΕ και DCIs ε, δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό. Οι κανονισμοί είναι πάρα πολύ παρόμοιοι, όπως σας είπα. Δεν έχω δυσκολία να επανεξετάσω το, τα μοντέλα ΑΚΕ και Κοτονού. Οι επικεφαλείς των μονάδων έχουν επιστρέψει από αντιπροσωπείες ε, στις οποίες δεν μπορέσαμε να δώσουμε, να αναθέσουμε θέσεις ε, διαχειριστών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ τα μάλα. Έχουμε τρεις ακόμα οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Ένα λεπτό την ερώτηση. Μια ερώτηση μπορείτε να τη θέσετε σε ένα λεπτό, αλλά όχι δύο. Ο κύριος ε, Τιάδης θα σας απαντήσει και θα ψηφίσουμε. Κύριε Στρίπερ, για σας Μία πάρα πολύ σύντομη ερώτηση. Βλέπω ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα σε θέματα συνεργασίας των κρατών μελών που γίνεται στην πράξη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για όλα αυτά τα επιμέρους μέτρα που αναφέρατε. Κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ να ευχηθώ να δουλέψει το νέο οργανόγραμμα της έκθεσης. Ωστόσο θα ήθελα να επεκταθώ λίγο στην ερώτηση του κυρίου Γκέρενς ίσως δεν έγιναν αντιληπτές όλες οι παράμετροι ή η επέκταση που θα μπορούσε να έχει και να ρωτήσω αν η κυρία Άστον θα μπορούσε να χειριστεί όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν μέσα από μια γενικευμένη πολιτική την ίδια στιγμή που θα μπορούσαμε με μια ανεξάρτητη επιτροπή που να έχει, ε, μια ανεξάρτητη δύναμη που να έχει και την έξωθεν καλή μαρτυρία τη ουδετερότητος, να παρεμβαίνουμε σε ζητήματα άμεση ανθρωπιστική κρίση, όπου δεν θα έχει σημασία με ποιον από του δύο εμπλεκόμενου θα κινηθεί αυτή η δύναμη. Νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα τη Βόρεια Αφρικής δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ. Θα συνεχιστεί και θα έχουμε νέε αναφλέξει, νέε συγκρούσει και το πρόβλημα θα είναι συνεχέ. Άρα δεν μπορεί κάθε φορά να λέμε ότι η κυρία Άστον εκφράζει την τάδε πολιτική και εμείς θα πρέπει να κάνουμε εκτόσεις με τον τάδε τρόπο. Θα είναι μια ανεξάρτητη task force, humanitarian task force, η οποία θα κάνει πάντοτε τη δουλειά της χωρίς να έχει να κάνει κάτι με την πολιτική που θα ακολουθούμε. Νομίζω είναι σημαντικό. Ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρνς για να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ. <clears throat> Εδώ και μήνες εγώ επιμένω πάντα στην ανάγκη να υπάρξει μια διορθωτική ενίσχυση του πόλου ανάπτυξης μέσα στο θερμισμικό ε, πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Γι' αυτό διερμηνεύω και μια αίτηση της κοινωνίας των πολιτών για να μπορέσει η Κομισιόν να δώσει τον εαυτό της την απαραίτητη δυνατότητα διατύπωσης προγραμμάτων, εκταμίευσης και υγιούς ε, διαχείρισης. Όλα αυτά γίνονται από εσά πολύ καλά, αλλά αυτό το οποίο δεν υπάρχει είναι να υπάρχει δυνατότητα σκέψης σε κάποια απόσταση από την καθημερινή τεχνοκρατική διαχείριση να αντιμετωπίσουμε ορισμένα προβλήματα τα οποία είναι στοιχειώδη. Κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μεγάλος χορηγός έχει το κύρος και το ειδικό βάρος που χρειάζεται να έχει σε παγκοσμίο Νομίζω όχι. Δεύτερον, το θέμα και εδώ το θέμα τη Κίνα στην Αφρική παίζει κάποιο ρόλο σε όλα αυτά. Και επίση το θέμα του πώ 27 χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να γίνουν αντιληπτοί σε παγκόσμιο επίπεδο σαν μία μονάχα δύναμη. Αυτή τη στιγμή το μονοπόλιο της πρωτοβουλίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε θεσμικό επίπεδο στα χέρια της Παγκόσμιας Τράπεζας και αυτή όμως μπορεί να κάνει λάθος. Γιατί έχουμε λοιπόν αυτή την υπερβολική μετριοφροσύνη όταν έχουμε τόσο σημαντικά υλικά μέσα στην διάθεσή μας. Γιατί δεν έχουμε μία μονάδα προβληματισμού για να δούμε μήπως μπορούμε να κινηθούμε καλύτερα. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν απαραίτητο. Και απαγοητεύουμε από την τωρινή κατάσταση. Τε, τέρμα οι ερωτήσεις, αλλά παρόλα αυτά... Σας πεθυμίζω το ερώτημα της κυρίας Κέλλερ και δεν μας είπατε τώρα πόσες γυναίκες έχουν πάρει διευθυντικές θέσεις μετά από αυτήν την νέα αναδιάρθρωση. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, για το θέμα το οποίο θέσατε, δύο διευθυντές θα έχουμε. <clears throat> από εννέα, δύο διευθυντές από εννέα είναι γυναίκες. Πιο πολλές θα θέλαμε, αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε περισσότερες έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα αυτά και φυσικά έχουμε κάθε υποχρέωση να βελτιώσουμε την ισότητα των φύλων στα ύπατα αξιώματα. Σε επίπεδο αρχηγών επικεφαλής τμήματων έχουμε πολύ περισσότερες ε, γυναίκες και εκεί είναι μικρότερο το πρόβλημα. Αποτελεσματικό της ε, βοήθειας και πώς μπορούμε να πείσουμε τα κάτι μέλη να μιλούν με μία μονάχα φωνή. Αυτό είναι απλό ερώτημα αλλά πρέπει να βρούμε μια πολυπλοκή απάντηση. Προβληματιζόμαστε για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Μέσα στα πλαίσια μια γενικότητα προβληματικής. Και αυτό το κάνει η μονάδα Α3, η οποία προβληματίζεται και αναστοχάζεται για το πώς θα πρέπει να γίνεται ο κοινός προγραμματισμός με τα κράτη-μέλη και για το είδος των προτάσεων που θα πρέπει να καταθέτουμε προς τα κράτη-μέλη ώστε να εξασφαλίσουμε την επιτυχία του εγχείρηματο. Είμαι κάπως σκεπτικιστής για το εγχείρημα αυτό, διότι ενώ πριν από κάποια χρόνια τα κράτη-μέλη είχαν ανοιχτό πνεύμα και ήταν υποστηρικτικοί για τον κοινό προγραμματισμό, για τις συμφωνίες σε σχέση με την κατανομή των αρμοδιοτήτων και των έργων. Νιώθω να υπάρχει απώλεια πίεσης ατμού, διότι αυξάνονται τα προβλήματα του προπολογισμού στα κάτι μελη Όσο περισσοτερα κάτι κράτη-μέλη έχουν να αντιμετωπίσουν περικοπέ στον αναπτυξιακό του προπολογισμό και είναι υποχρεωμένοι να αποσυρθούν από χώρε και μέρη του κόσμου, λιγότερο ενθουσιασμό θα έχουν ω εκ τούτου και για τη συνεργασία μαζί μα αρνητικός συσχετισμός για τον οποίο εγώ ανησυχώ. Γι' αυτό θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις που θα ξαναφέρουν τις χώρες αυτές σε ένα κοινό εγχείρημα μαζί μας. <clears throat> Το γεγονός ότι δαπανούμε πολλά χρήματα αλλά δεν έχουμε την ορατότητα που θα έπρεπε να έχουμε είτε έναντι των άλλων χορηγών είτε άλλων μεγάλων χώρων στον κόσμο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και συμφωνώ και εγώ και καν να γνωρίζω <clears throat> ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε. Να έχουμε λοιπόν μια περαιτέρω ανάλυση των θέματων αυτών. Έχουμε την ικανότητα μιας ανθρωπιστικής α, ε, αντιμετώπισης ανεξάρτητα από από πολιτικές συγκυρίες. Αυτό είναι η υπηρεσία ΕΚΟ της Κομισιόν, η οποία παραμένει παρά την ύπαρξη υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ανεξάρτητη και αυτόνομη στην δράση της. Τώρα το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε συνεκτικότητα πολιτικής δράσης μας με την υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης. Αν θα μπορέσουμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό στον τομέα της ανάπτυξης, αυτό θα χρειαζόταν πολύ συζήτηση και καταλαβαίνω θέλετε να ψηφίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε και την απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Μπορούμε μέχρι και να σας χειροκροτήσουμε. Δύο λεπτά για να τακτοποιηθούμε και να περάσουμε στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Πάτε τις κάρτες σας παρακαλώ.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 Voilà, nous allons procéder à un essai. Alors. Να κάνουμε μια δοκιμή. Ψηφίστε όλοι παρακαλώ. Σας θέτω ένα ερώτημα. Καθυστερήσαμε, ναι ή όχι. Ψηφίστε ναι ή όχι. Ή και αποχή μπορείτε να κάνετε. Ça marche Alors pour le moment, on n'est pas encore Εντάξει, μια χαρά είναι τα πράγματα προς στιγμή. 26, 17, 18 έχουν ψηφίσει, 19, ναι έρχονται, έρχονται. Εντάξει, και εγώ ψήφισα. Τρεις δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Άλλοι δύο έχουν μείνει, ένα άτομο δεν έχει ψηφίσει. Ένα άτομο λείπει. Μήπως έχει καθυστερήσει. Oui, Εκτός αν έχουμε τεχνικό πρόβλημα. Ah, Ωραία. Ε, το δικό μου μαραφέτη δεν δούλευε. Euh, euh, να σας υπενθυμίσω καταρχήν ότι υπάρχει μια μικρή διόρθωση στον κατάλογο ψηφοφορία για την παράγραφο 8. Η τροπολογία 67 είναι... Έχει εκπέσει αν εγκριθεί η τροπολογία 66, όχι 65. Θέλετε να τα ξαναπώ αυτά. Παράγραφος 8 η 67 εκπίπτει, αν εγκριθεί η 66 και ουχή η 65 ως εσφαλμένος γράφει ο κατάλογος της ψηφοφορίας. Εντάξει. Θα ξεκινήσω. Η έκθεση Κάσμαρεκ είναι το πρώτο έγγραφο που θα ψηφίσουμε. Πρόβλημα. Nous allons Alors, amendement... Τροπολογία 9. Ηλεκτρονικά θα τα κάνουμε όλα. Α, διανατάσσεως χειρών. Μου είπαν ότι όλα ηλεκτρικά πρέπει να γίνονται, όχι. Α, αλλάζουν τα πάντα τότε. Αλλάζουν τα πάντα, λέει η πρόεδρος. Διανατάσσεως. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική β υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 21. Στην παράγραφο 2. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έλεγχος, έλεγχος. Για την 23 ψήφι άρχεται η ψηφοφορία. εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ <clears throat> κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές <clears throat> εγκρίνεται τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 στην παράγραφο 4 ψήφι υπέρ 37. κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το δεύτερο τμήμα Δεύτερο τμήμα της 40 ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία προφορική υπαριθμών 1 Μακλάρκιν. Κυρία Κλάρκιν, συγγνώμη, τι είναι αυτά που λέω. Υπέρ. Κατά. Αποχέ <clears throat> θα ελέγξουμε. Προφορική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές δεχτή 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 έχει 51 έχει πέσει εκπέσει τουλάχιστον Συμβιβαστική εύση μετά στα ελληνικά, <clears throat> ψήφι υπέρ, πρώτο τμήμα, συγγνώμη, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, ε, έλεγχος. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 52. Μόνο το δεύτερο τμήμα της 52. 52 δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 54, όχι, όχι, 54. 57, 57. 53. υπέρ, κατά, Εφόσον ενεκρίθη 52, ναι, αλλά η λέξη αν το πείτε στο μικρόφωνο θα καταλάβουμε, γιατί εγώ στα αγγλικά δεν ξέρω πώς να τα πω αυτά. Εάν έχει εκριθεί η F, κάτι το οποίο είναι γνωστό ότι έγινε, η λέξη particular, li πρέπει να γίνει and also. Αυτό είναι η τροπολογία. Ωραία τα είπατε. Αν τα λέγω εγώ στα αγγλικά θα καταλαβαίνετε μία. Λοιπόν, τροπολογία 53, ψήφι υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Δεν <clears throat> 57 υπέρ. Κατά. Όχι. Δεκτή. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική G. G αγγλικά. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ξέρετε δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή 69 έχει εκπέσει παράγραφος 9 συμβαστική H ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 70 όχι 74 υπέρ Κατά. Αποχές ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote Πέρας. Ποιος δεν ψήφισε. Εγκρίνεται. 75. Εκπίπτει. 77 ψήφι υπέρ. Κατά. Την 76 την ξεχάσατε. Συγγνώμη. Εβδομήντα Συγγνώμη. Πρώτο τμήμα. Ψήφι περ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 79 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 79 ηλεκτρονικά άρχεται γρήγορα πέρας απογείδεται παράφος 10 προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 82 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την 82 πέρας Δεκτή. Προφορική 3 υπέρ. Κατά. έτσι δεκτή. 83. Εκπίπτει 83. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Εποχές. δεκτή. Ο, συνεχίζουμε. 88. υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 89 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 90 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 91 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά. Ελέγχουμε για την 92 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 93 υπέρ. Κατά. Από χε δεκτή. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Θα δούμε. Θα ελέγξουμε. Έχουν κουραστεί τα χέρια σας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική δε υπέρ. Κατά δεκτή. Συνεχίζουμε με την 104 για την παράγραφο 13. 104. Όχι, δεν τη θέλετε. Ναι, ναι. 104 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 5 <clears throat> υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Εκπίπτει 107. Πάμε στην 108 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται κρίμα. Να το ελέγξουμε. Έλεγχος για την 109. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Με μία ψήφο μονάχα. 111 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική J υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 113 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 115 υπέρ <clears throat> κατά αποχές δεκτή. 100 και 117 συνεπαρασύρθη. 117 εκπίπτει αν απορρίπτεται η 116. Ή εάν εκπέσει βέβαια. Μπράβο αν. Μπράβο αν. Μπράβο. Πού είμαστε. 118. Υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Ή ίσως εγκρίνεται. Έλεγχος για την 118. Άρχεται η ψηφοφορία στην 118. Πέρας. Ε, εγκρίνεται. Ε, δεν, δεν σηκώσατε καλά τα χέρια σας. 119 υπέρ κατά. Απόχες εγκρίνεται. 120 όμως 100 υπέρ κατά. Απόχε απορρίπτεται. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 16, συμβιβαστική κάπα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 124 παράγραφος 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. 125 με 128 μπλοκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Παράγραφος 17 συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος... Όχι. Προφορική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 17, τοπολογία 134, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 134. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρα, παράγραφος 18, 135 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 141. Πέρας. Εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικός άρχεται η ψηφοφορία για την 146 πέρας εγκρίνεται Παράγραφος 19, συμβιβαστική M, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 147 149, παράγραφος 19. Όχι. Ο κύριος Κάσμαν, δεν νομίζω ότι 145 εγκρίθηκε. Άρα πού είμαστε. Καταπίπτει μόνο αν εγκριθεί 145. Η, 100... η 145 όμως απορρίφθηκε. Άρα έχετε δίκιο, κύριε Κάσμαν είδατε τη η βοηθή μου. Όλο λάθη κάνουν. 148 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 19. 150 τροπολογία, δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα τη 150. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20. Συμβιβαστική εν υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 100... Διορθώνει πρόεδρος. Ε, στην 151 είμαστε. Μην τσεκώνεστε μεταξύ σας. 157 τότε, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 21, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συγγνώμη, είχα ξεχάσει ότι είναι η συμβιβαστική O, αλλά νομίζω ότι εντάξει, καταλάβατε. Άρα φτάνουμε τώρα στην 163. Διαφωνούν εδώ οι βοηθοί μου. Anne-Louise qui a besoin de chocolat. 162. Λοιπόν, 162, υπέρ. Ευχαριστώ. Καταπίπτει αν εγκριθεί 163 Άρα η 168. Αλλά η 168, άρα 162. Συμφωνείτε? Είμαστε τρεις εδώ πέρα. 162. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Έναρξη ψηφοφορίας για την 162. Πέρας. Εγκρίνεται. 161. Ε, εκπίπτει, ε, ή δεν εκπίπτει. 161, πάση περιπτώσει. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20, ε, παράγραφος 21, τροπολογία 163, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 164, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Έναρξη για την 165. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 21. Τροπολογία 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Παράγραφος 22, συμβιβασμός π σε δύο μέρη. Υπέρ του πρώτου μέρους. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Δεύτερο μέρος του συμβιβασμού π Έναρξη. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 22, τροπολογία 172, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι είναι υπέρ, ναι, ναι, εγκρίνεται. Παράγραφος 23, συμβιβασμός R, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. εκατόν εκατόν εβδομήντα τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εκατόν εβδομήντα έξι εκπίπτει 20, παράγραφος 23, 178 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 23, η 179 και η 180, και μαζί. Πρώτο μέρος, παρά τα αυτά υπάρχουν μέρη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Οι τρεις ε, μαζί, όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, η 181 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 185 Παράγραφος 23, 185 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 23, τροπολογία 186 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 187 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 188 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η ιδεολογική σκέψη Β, η 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται έχασα τα λόγια μου λέει η πρόεδρος αιτιολογική σκέψη σε ε, τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η ε, παράθεση 4 τροπολογία 1 Λοιπόν, οι τέσσερις πρώτες μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με την προφορική τροπολογία εδώ. Λοιπόν, φτάνουμε στην τροπολογία παριθμών 4, 5 με συγχωρείτε λέει πρόεδρος. Η, η πέντε καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε η τρία. Σύμφωνοι. Άρα φτάσαμε στην έξι. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οπότε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τελική ψηφοφορία, έναρξη, πέρας, εγκρίνεται. Ορίστε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Οπότε θα περάσουμε στο επόμενο. Κύριο Τιβάς,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 Θα ξεκινήσουμε με την παράγραφο 1, τροπολογία 18, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21, παράγραφος 4, 21, σε δύο μέρη, πρώτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση την 26. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 6, τροπολογία 27, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 28, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30, υπέρ. Όχι, όχι, όχι, όχι. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία προφορική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 33, παράγραφος 12, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 13, τροπολογία 34 σε δύο μέρη, υπέρ, 34 λοιπόν σε δύο μέρη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο μέρος εκπίπτει έλεγχος έλεγχος πρώτο μέρος έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας πέρας εγκρίνεται Εγκρίνεται. Πολύ καλά κάνατε και ζητήσατε έλεγχο. Οπότε ψηφίσουμε το δεύτερο μέρος. Υπέρ. Σηκώστε το χέρι σας ψηλά σας παρακαλώ. Έχει επέλθει κόποση αλλά σηκώστε το χέρι σας. Ευτυχώς που είσαστε εδώ στην πρώτη σειρά γιατί δεν το σηκώνετε ψηλά. Να ορίστε. Κατά. Ε, να κατεβάσετε το βλέμμα Εν περιπτώσει. Λοιπόν, ξεκινάμε το δεύτερο μέρος. Ζητώ συγγνώμη κύριε Γκρίνς. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Όχι. Απορρίπτεται. Χωριστή ψηφοφορία. Στην αρχική παράγραφο 13, χωριστή ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος είναι η δεύτερη προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, ησυχία σας παρακαλώ μην μιλάτε μεταξύ σας. Εγκρίνεται τώρα η 35 εκπίπτει, η 36 σε τρία μέρη. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, επαλήθευση. Για το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 36, έναρξη, πέρας, απορρίπτεται. Τρίτο μέρος, υπέρ, κατά, επαλήθευση. Το τρίτο μέρος το επαληθεύουμε, έναρξη, πέρας, Απορρίπτεται. Παράγραφος 14, τροπολογή 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 14 ή 38 σε δύο μέρη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά επαλήθευση του δεύτερου μέρους στις 38 έναρξη. Πέρας Απορρίπτεται. Παράγραφος 15, τροπολογία 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει ε, η 41 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 42 υπέρ. Κατά σε δύο μέρη, αν δεν είχα δει το δεύτερο μέρος, λοιπόν, σε δύο μέρη. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 15, η 43 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται με τα τσαρούχια λέει η πρόεδρος εδώ γίνεται καυγά στη γραμματεία λέει η πρόεδρος απορρίφθηκε όμως 46 υπέρ κατά Ελέγχουμε τη 46. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Χωριστή ψηφοφορία για την παράγραφο 16. Παρακαλώ. Είπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται, εγκρίνεται, είπα εγκρίνεται, εγκρίνεται. Καλά, ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα της 49. Πέρασε εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε θα ελέγξουμε ελέγξουμε για την 54 ηλεκτρονικά πέρας απορρίφθηκε χωριστή ψηφοφορία για την παράγραφο 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία στην 56 Πέρασε. Εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ υπέρ κατά αποχές έλεγχος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 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ σε τμήματα, σε τμήματα, συγγνώμη. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τρία. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 ως 17 από κοινού αν συμφωνείτε. 13 με 17. 13 με 17. Ακούστε με, 13 με 17 όλες μαζί, υπέρ, κατά, αποχές δεκτές. Αιτιολογικές αναφορές. Από κοινού, όλες μαζί, μέχρι τις θέσεις, όλες μαζί, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Μία μικρή ανακοινωσούλα για την επόμενη ψηφοφορία η Γραμματεία έχει διανύμει ένα κατάλογο με προφορικές τροπολογίες του ΕΛΚ για τις εξής τροπολογίες 5, 11, 38 και 59. Ο κ. Μητσέα δεν παρόν. Κανονικά θα έπρεπε ο, ο εισηγητής να τις παρουσιάσει. Κύριε Σφένσον θα πάτε εσείς το λόγο. Θα τις διαβάσει ο κ. Σφένσον. C'est un français, quand même. S'il vous plaît, faites un peu moins de bruit, parce qu'on va continuer. Λίγο λιγότερο θόρυβο. Είναι δύσκολο όταν κουβεντιάζετε όλοι. Πάμε να τα κάνουμε όλα πιο γρήγορα. Πιο... Μπορούμε, εντάξει, πάμε. Γκέρενς. Παράγραφος 1, τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Οπότε. Περνάμε στην ΑΦΕΤ τροπολογία 1 παράγραφος 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είστε έτοιμοι? Ωραία. Τον προπολογισμό είναι 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αφέτ 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμό 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αφέτ 13. Τρία τμήματα. Υπέρ. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Έλεγχο ηλεκτρονικός της ΑΦΕΤ 13 στο δεύτερο τμήμα έναρξη ψηφοφορία. πέρας απορρίπτεται περνάμε στο τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε τότε ηλεκτρονικά το τρίτο τμήμα της ΑΦΕΤ 13, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Ωραία. Άλλα τα χέρια, άλλα γράφουν οι οθόνες. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικτός. Έναρξη της ε, ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 24. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25 παράγραφος 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 26 καταπίπτει άρα 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Κύριε Γκέρνς, θέλετε να πάρετε το λόγο μετά την 29 από ό,τι κατάλαβα. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην 29. 28 τότε ψηφίζουμε. Υπέρ. Α, είναι και για άλλη έκθεση. Λοιπόν, τροπολογία 28, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Έναρξη ψηφοφορίας για την 28. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχο Ή όχι. Εντάξει, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Την 30. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφο 3. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όλα τα υπόλοιπα καταπίπτουν θα ψηφίσουμε τον προπολογισμό την τροπολογία 4. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρα, να δώσω το λόγο στον κύριο Σφένσον για την παράγραφο 4. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. κυρία Πρόεδρε. Εμείς θέλουμε να συμπεριλάβουμε το ότι ο δημοκρατικός δημοσιονομικός έλεγχος τη χώρες Δικαιούχου θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δημοσιονομική υποστήριξη και ζητά επίσης ευρεία συμμετοχή των κοινοβουλίων και την διαβούλευση με την, με την κοινωνία των πολιτών στις χώρες εταίρου για να αποφασιστεί δημοκρατικά η χρήση των ε, δημοσιονομικών κονδυλίων. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά θέλαμε να προσθεθούν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία. Κοντ 2. Υπέρ. Κατά. Δεν παρακολουθείτε όλοι. Θα πρέπει να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Κοντ 2. Παράγραφος 4α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κόντ 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική παριθμών 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τότε στην ΑΦΕΤ 6. Παράγραφος 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μήπως μπορείτε να κάνετε ησυχία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι να παρακολουθήσουμε. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40... Όχι 44. 44 και μετά όλες μαζί τις υπόλοιπες πρωτοπολογίες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, όλες μαζί από τις 46, από τις 45 συγγνώμη λέει η Πρόεδρος, μέχρι τις 47. Ωραία. 45 με 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκρίνονται. Αφέτ 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 49 καταπίπτει. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κοντ 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αφέτ 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 51 καταπίπτει. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μπιτζ 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κόντ 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κόντ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κόντ 9 παράγραφος 8 δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Παράγραφος 8, bridge 6, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Αφέτο 8 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικός έναρξη ηλεκτρονική ψηφοφορία για την Αφέτο 8 πέρας εγκρίνεται Παράγραφος 10, 57 τροπολογία. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αφέτε 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη προφορική τροπολογία. Κύριε Σφένσον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε πιστεύει ότι οι χώρες που είναι πλούσια πετρέλαιο και μεταλλεύματα έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τη δική τους ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας μέσω διαφανών συστημάτων συλλογή φόρων και την σωστή κατανομή του πλούτου. Ζητεί λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό ω ζήτημα προτεραιότητα προκειμένου να, στα... να καταργηθεί σταδιακά η δημοσιονομική στήριξη. Ευχαριστώ. Υπέρ. Κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς ε, την προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 59 καταπίπτει. Άρα πάμε στην 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αφέτ. Α, όχι, δεν πάμε εκεί. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αφέτ 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Κοντ 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αφέτ 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αφέτ 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικό στην 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Bridge 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Bridge 11. Τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικό στο τρίτο τμήμα της Bridge 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται, αλλά ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς το τέταρτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ωραία, παράγραφος 15, τροπολογία 68 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Bridge 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Bridge 13, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κύριε Σβένσον, έχετε το λόγο για την προφορική τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όταν ε, η δημοσιονομική στήριξη είναι βασική μορφή ενίσχυσης και όταν είναι στόχος ε, να έχει στόχο να ενισχύσει την δημοσιονομική αυτή στήριξη κατά τα επόμενα έτη και συνεχίζει το κείμενο. Θέλουμε να διαγραφούν όμως οι υπογραμμισμένες, ε, το υπογραμμισμένο τμήμα της φράσης. Δηλαδή το κομμάτι and whereas μέχρι το coming years. Να το διαγράψουμε θέλουμε αυτό. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικό στην προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρα πάμε στην τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Κύριε Γκέρενς, με κοιτάτε και γελάτε και με αποσταθεροποιηθεί. Δεν μπορώ να παραμείνω σοβαρή. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη για το αποτέλεσμα, οπότε να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 6. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Πάω πάρα πολύ γρήγορα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνω μερικέ παύσει γιατί τα χάνω. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία τελευταία, κύριε Βένσον, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε να συμπεριλάβουμε τις εξή λέξεις. Ε, όταν η δημοσιονομική στήριξη βοηθά στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας ενίσχυσης ε, βάσει των αρχών της κυριότητας και της εναρμόνισης, ε, δεδομένου του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των δωρητών και των δικαιούχων, καθιστά δυνατή την προσαρμογή των συνεισφορών ε, στις χώρες προτεραιότητας, όταν έχουν συμπεριληφθεί οι προσαρμογές αυτές στις ε, στα εθνικές στρατηγικές ε, για την καταπολέμηση της φτώχειας. Θέλουμε να, το should, να συμπεριληφθεί το should help, όπως σας διάβασα. Λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ. Καταπίπτει. Λάθος. Πάμε τώρα σε αιτιολογικές αναφορές. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Δεν σηκώσατε καλά τα χεράκια. Θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς τότε. Άρα, Έναρξη ψηφοφορία για την τροπολογία 3. Πέρα. Απορρίπτεται. Τώρα θα κάνουμε την τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έχουμε μία τελευταία ψηφοφορία. Ah, je suis en train de la hmm euh, oui. Alors, nous allons bien. Λοιπόν, θα κλείσουμε με την έκθεση του κυρίου Γκέρενς. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Παράγραφος 1, τροπολογία 2, υπέρ. Γεια σας. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 1. Συμβασμός 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παραγραφο. Συμβιβασμός 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφ, ε, τροπολογία 7 με συγχωρείτε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3 σε δύο μέρη. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο μέρος υπέρ κατά α, πρόβλημα δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές επαλήθευση δεύτερο μέρος του συμβιβασμού 3 επαλήθευση έναρξη πέρας εγκρίνεται τροπολογία 11 ή 16. Τι λέτε. 16. Παράγραφος 5, τροπολογία 16. Υπέρ. Κύριε Γκέρενς, είστε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παρά, ε, τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Ευχαριστώ κύριε Γκέρενς. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Αποχές. Δεν είμαι σίγουρη να ελέγξουμε τη 19 έναρξη πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 20, 22, 22 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 και 25 και 26 υπέρ των τριών αυτών κατά αποχές εγκρίνονται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική του κύριου Γκέρενς. Ζητήσατε το λόγο κύριε Γκέρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το εξή κείμενο. Θέλω να αντικαταστήσω το κείμενο από αυτό που θα σας διαβάζω. Θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο πρώτος πάροχος κονδυλίων που σκοπό έχουν ε, την ανάπτυξη πρέπει να πάρει την ηγετική θέση σε θέματα ανάπτυξης και θεωρεί ότι πρέπει μία εσωτερική ανεξάρτητη μονάδα να βοηθά την Κομισιόν στις πολιτικές επιλογές της. Ο κύριος Μπέργμαν διαφωνεί. δεν, του πήγαν καλά τα πράγματα, γι' αυτό λέει ο κύριος Γκέρνς. Θα ψηφίσω, αλλά είμαι κατά. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ αυτής της προφορικής τροπολογίας. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Je euh, Λοιπόν, σας επιτρέπω να βγείτε από την αίθουσα με ησυχία ε, για τρία λεπτά και παρακαλώ σεβασμό σε αυτούς που συνεχίζουν τη συνεδρία. Λοιπόν, σε λίγο θα ξεκινήσουμε. Σας παρακαλώ, καθίστε. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε. Έχουμε μισή ώρα καθυστέρηση. Σα Σας ευχαριστούμε όλες. Οι άντρες δεν μετράνε. Καθίστε παρακαλώ. Δεν ξέρω τώρα πού βρίσκονται οι ομάδες επισκεπτών. Δεν έχετε θέση στα έδρανα πίσω. Όλοι αυτοί που έχουν ε, ρέγκλες παρακαλώ να καθίσουν. Οι ομαδες επισκεπτων δεν εχετε θεση στα εδρα να πισω ολοι αυτοι που εχουν ρεγλες παρακαλω να καθισουν οι υπολοιπες παρακαλω Έχω την μεγάλη τιμή και χαρά να χαιρετήσω την κυρία Εύα Μπριτ Σβένσον, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και της Ισότητας των Φίλων και όλα τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών για το γεγονός ότι είναι παρούσες στη συνεδρίασή μας. Σήμερα θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της σεξουαλικής βίας στις ένοπλες συγκρούσεις με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση στη δημοκρατική δημοκρατία του Κονγκό. Έχουμε προσκαλέσει και την κυρία Μαργό Γουόλστρομ, πρώην επίτροπο και τώρα ειδική εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία στι ένοπλε συγκρούσει και τον ε, ε, ιατρό Μουσβέκ, ο οποίο είναι γιατρό στον Μπουκάβο και ε, επίσης βραβείο Ρουά Μποντουέν για την ανάπτυξη 2010-2011 που του απενεμήθη χθες στις Παρακαλώ, παρακαλώ. Και χαιρετίζω την παρουσία του κυρίου Ρίμποβα Σάκανη, συγγνώμη για την ε, προφορά μου, ο οποίος είναι ο πρεσβευτής της Δημοκρατικής Δημοκρατίας του Κονγκό και επίσης είναι παρόν του εκπροσώπου του πρέσβεως του Κονγκό. Σα υπενθυμίζω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα αντιμετωπίσει το θέμα αυτό και έχει εγκρίνει ψηφίσματα που καταδικάζουν τι πράξει που έχουν λάβει η χώρα. Οι δύο επιτροπέ μα θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μία, μία επικέντρωση στα θέματα αυτά τη κοινή γνώμη και θεωρούμε ότι η πείρα των δύο προσωπικότητων που είναι προσκεκλημένοι μας, που αγωνίζονται κατά αυτού, αυτής της μάστιγος από διαφορετικές οπτικές γωνίες, είναι πολύ χρήσιμο για το κοινοβούλιο. Δίνω καταρχήν το λόγο για την κυρία Βόλστον κατά 20 λεπτά ή 15, αν μπορεί τουλάχιστον, για να απολάβουμε. για να μας παρουσιάσει το έργο της στα Ηνωμένα Έθνη και τις επιτυχίες που έχει καταγάγει μέχρι στιγμής αλλά και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Μικβέγ για να μας εξηγήσει τη δική του επιτόπια εμπειρία. Πρώτα η κυρία Γόλστομ για 15 με 20 λεπτά. Έχετε το λόγο, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για μένα να είμαι πάλι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βέβαια με άλλη ιδιότητα, για να αναφερθώ σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να είμαι μαζί με τον δόκτωρα Μουκ ο οποίος είναι γνωστός σε όλους σας τώρα από το έργο του στο Μπουκάβου και θέλω να εξασφαλίσω ότι και αυτός θα έχει αρκετό χρόνο για να απαντήσει τα ερωτήματά σας και να σας δώσει και τις δικές του απόψεις. Εγώ έχω τώρα μια τελείως νέα θέση στα Ηνωμένα Έθνη που δημιουργήθηκε πριν από ένα έτος βάσει ενός από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που αντιμετωπίζει το θέμα των γυναικών, τη ειρήνη και τη ασφάλεια. Μας χειρίζει 10 χρόνια στο παρελθόν όταν έτυχε αναγνώριση το γεγονό ότι ο πόλεμο και η ειρήνη επηρεάζουν διαφορετικά του άνδρες και τι γυναίκε. Και οι γυναίκε θα πρέπει να έχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσουν στι διαπραγματεύσει για ειρήνευση. Σε πρόσφατα, πρόσφατα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφάλεια αντιμετωπίζει και το θέμα τη σεξουαλική βία ω όπλου πολέμου και έτυχε αναγνώσει βάσει του ψηφίσματο που θέσπισε τη θέση μου, αποφασίστηκε ότι τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την παγκόσμια μάστιγα. Δεν είναι ένα θέμα μονάχα που αφορά το Κονγκό ή την Αφρική, αλλά είναι κάτι το οποίο σοβεί σε όλους σχεδόν του πολέμους και τι ένοπλε συγκρούσει σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ατιμορρησία, να την τερματίσουμε να κινητοποιήσουμε την πολιτική ηγεσία, να εξασφαλίσουμε ότι ο ΙΕ και η διεθνή κοινότητα μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στα προβλήματα αυτά και φυσικά πρέπει να δώσουμε στι γυναίκε τη δυνατότητα συμμετοχή μέσω των πολιτικών μα για να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκε έχουν μια φωνή και συμμετέχουν στι λήψει αποφάσεων. Όπω είπα, ο ρόλο μου είναι παγκόσμιο, Αυτό σημαίνει ότι εγώ και η ομάδα μου, η μικρή μου ομάδα, είμαστε νέα άτομα συνολικά. Έχουμε να δράσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε 7 χώρε στι οποίε εστιαζόμαστε. Μία από αυτέ είναι το Κονγκό. Υπάρχουν άλλε 4 στην Αφρική, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Σουδάν, το σύνολο του Σουδάν αυτή τη στιγμή, πριν από τον διχασμό του, η ακτή ελεφαντοστού, επίσης Βοσνία Ζεγοβίνη στην Ευρώπη και Κολομβία εκτός της Αφρικής. Χώρες όπου υπάρχουν ακόμα προβλήματα και υπάρχει και πρόβλημα απόδοσης δικαιοσύνης για τα θύματα σεξουαλικής βίας. Δύο λέξεις όταν συζητούμε για αυτό το φαινόμενο σε ιστορικό βάθος. Ορισμένοι λένε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδύρυτο, ότι πρέπει να θεωρηθεί παράπλευρη ζημία του πολέμου είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να αποφύγει σε συγκρούσεις και σε πολέμους. Μια άλλη έκφραση είναι ότι είναι κάτι το οποίο δεν αναφέρεται ποτέ. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λεχθεί. Ακόμα και στη δίκη της Νιρεβέργης δεν περιγράφησαν αυτές οι ομότητες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν και τα δύο αυτά θέματα. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι κάτι απαραίτητο. Ο μαζικός βιασμός δεν είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο ή αδύνητο ούτε και η μαζική φόνη. Ε, μαζική Και αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε ούτε να το συγχωρήσουμε. Πρέπει αντίθετα να το καταδικάζουμε με όλες τις πολιτικές μας πράξεις. Και επίσης πρέπει να δοθεί φωνή στα θύματα. Πρέπει το θέμα αυτό να έρθει στην επικαιρότητα, να μην παραμείνει, στην, ε, να μην παραμείνει ένα βοβό πρόβλημα, ένα βοβό βάσανο. Πρέπει λοιπόν να Μιλάμε για αυτό το θέμα και αυτό πρέπει να κάνουμε πάντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά τα θέματα που κάνετε πρέπει να θέτουν το ερώτημα τι γίνεται σε αυτές τις συγκρούσεις. Εάν δεν συζητά κανείς για αυτό το θέμα, δεν θα ξέρουμε ποτέ ποια είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να ενσωματωθεί λοιπόν σε όλες τις πολιτικές μας. Ένα ακόμα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Στην Δημοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό αυτό που κρατάει τις συγκρούσεις αυτές ζωντανές, αυτό που χρηματοδοτεί τη δράση των ενόπλων ομάδων, είναι οι εξορρυκτικές δραστηριότητες. Γι' αυτό όλες αυτές οι συγκρούσεις για τα ορυκτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν εγκρίνει ήδη νομοθεσία που λέει ότι θα πρέπει να χαρτογραφήσουμε όλες αυτές τις ε, διαδικασίες συγκρούσεων και να ανοιχνεύσουμε την προέλευση των ορυκτών πόρων που έρχονται από τις χώρες αυτές. Ελπίζω ότι μαζί με τις ΗΠΑ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να καταλήξει ένα κοινό καθεστώ όπως αυτό και για τα διαμάντια που προέρχονται από ζώνες συγκρούσεων. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχει μια πρωτοβουλία για τα θέματα αυτά και όπως είπαμε το πρόσφατο ψήφισμα το 1960 του προηγούμενου Δεκεμβρίου έχουμε πια πρόσβαση σε όλη την εργαλειοθήκη του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο σημαίνει ότι από εδώ και πέρα μπορούμε να παρακολουθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό το πρόβλημα και να εκδίδουμε εκθέσεις για όλα αυτά. Για να έχουμε λοιπόν καλύτερα στοιχεία στο βαθμό του δυνατού, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλο όνειδος και στιγματισμός για αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή για κάθε έγκλημα, για κάθε αδίκημα το οποίο έρχεται στη δημοσιότητα μπορεί να είναι άλλα 50 αντίστοιχα τα οποία μένουν κρυφά και πρέπει να μπορούμε να κατονομάσουμε και να επωνυδίσουμε αυτούς οι οποίοι διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα. Πρέπει επίσης να έχουμε πρόσβαση στις κυρώσεις που είναι στη διάθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δηλαδή πάγωμα στοιχείων ενεργητικού, απαγόρευση ταξιδίου ή προξενικής θεώρησης για τους δράστες. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για να μπορέσει να σταματήσει η ατιμορρησία. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι στι διαπραγματεύσει ειρήνη θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια γυναίκα στις διαπραγματεύσεις. Σε 300 συμφωνίες που έχουν γίνει για τα θέματα ειρήνευση την τελευταία δεκαετία, ε, δεκαετία μόνο, 18, μόνο σε 18 από αυτές τις διαδικασίες αναφέρθηκε η σεξουαλική βία. Αυτό είναι μόνο η κορφή του παγόβουνου. Αν δεν υπάρχουν γυναίκες στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, τότε ουσιαστικά αγνοούμε το ίμιση του πληθυσμού σε αυτές τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την ειρήνη και την ασφάλεια. Εξακολουθούμε λοιπόν να υποτιμούμε τον πραγματικό αντίκτυπο της σεξουαλικής βίας που υφίστανται τόσες πολλές γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα πραγματικό εμπόδιο στην επίτευξη της ειρήνης και της ασφάλειας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Έχουμε δει μονάχα την εκκίνηση αυτών των προβλημάτων, τα οποία στη συνέχεια κρατάνε για γενιές. Η οποιαδήποτε προσπάθεια επίτευξης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στη συνέχεια είναι πολύ πιο δύσκολη, είναι υποθηκευμένη, είναι πιο δύσκολη και για την διεθνή κοινότητα εάν δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό και φυσικά τα βάσανα αυτών των γυναικών δεν έχουν τέλος. Ό,τι κάνετε λοιπόν στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά θα πρέπει να προσπαθήσετε να εξασφαλίσετε ότι θα πρέπει να σπάσει το ταμπού τη σιωπή, θα πρέπει να τεθούν τα ερωτήματα, θα πρέπει τα θέματα αυτά να αναφέρονται εκπεφρασμένα. Το τελευταίο παράδειγμα είναι η Λιβύη γιατί παρά το γεγονό ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας πέρασε ένα φιλόδοξο ψήφισμα, δεν είπε τίποτα για τη σεξουαλική βία, ιδίω στα ψηφίσματα αυτά 1970-1973 για την Λιβύη, ενώ ξέρουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Στη Δημοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό αυτό εξακολουθεί να είναι η Λιβύη αλήθως των προσπαθειών μας. Και επίσης της διεθνούς αλληλεγγύης μας δηλαδή το πόσο αποφασιστικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και όλα ξεκινούν με το σπάσιμο της σιωπής. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε, ευχαριστώ που θέτετε στην επικαιρότητα το θέμα αυτό και στο προσκήνιο και συζητάτε μαζί μας <clears throat> και η ελπίδα μου είναι ότι θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ ΗΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα και θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μάστιγα. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Euh, Δίνω το λόγο στον ε, δόκτωρα Μουκβέγγι. 15 με 20 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Μετά την ε, παρουσίαση ε, της κυρίας Μάργοτ Βάλμστρομ για, την, ε, για, τους, για τους βιασμούς. Θα ήθελα να σας πω ότι η κατάσταση που είναι στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό παρατηρείται εδώ και 15 χρόνια. Θα ήθελα να πω ότι οι βιασμοί που γίνονται στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, σε αντίθεση με αυτό που μερικές φορές ακούμε από τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι ένα πολιτιστικό γεγονός, είναι μια συνέπεια του πολέμου και νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώς η ένοπλη σύραξη μπορεί μεν να εξελίσσεται, αλλά και τα εγκλήματα που γίνονται κατά τη διάρκεια της περίοδου της σύγκρουσης, αλλά και μετά τη σύγκρουση, δίνουν τη δυνατότητα ύπαρξη τέτοιου είδους εγκλημάτων, όπως οι βιασμοί για παράδειγμα. Πρόκειται για ένα έγκλημα που ε, γίνεται στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, το έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές, είναι συστηματικής φύσεως ε, και όταν λέω συστηματικής εννοώ ότι αφορά ολόκληρα χωριά και δεν μιλάω τώρα για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, ε, ούτε για συγκεκριμένα φύλακαν των ανθρώπων που είναι θύματα βιασμού στα συγκεκριμένα χωριά. Οι ομάδες που κάνουν τους βιασμούς αυτούς έχουν συγκεκριμένες μεθόδους και οι μέθοδοι αυτοί είναι πολλές φορές... Ε, δεν ε, είναι πάρα πολύ εμφανής αν μια ομάδα μπορεί να διαπράξει βιασμό με μεθοδικό τρόπο, με μια μέθοδο ε, κάπως συγκεκριμένη, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε κάπως να εντοπίσουμε αυτή την ομάδα και αυτό σημαίνει ότι είναι, σχεδιασμένες, είναι προσχεδιασμένα αυτά τα εγκλήματα. Αν είναι προσχεδιασμένα, πρέπει να υπάρχει και ένα κίνητρο. Το κίνητρο, λοιπόν, που ε, υπάρχει και η ε, κυρία Μάλμστρομ το είπε ήδη, είναι η πρόθεση εκμετάλλευσης ε, παρανόμως ε, των ε, φυσικών πόρων της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό. Όμως για να γίνει αυτή η παράνομη εκμετάλλευση ο στόχος είναι να φύγει, να εκδιωχθεί ο πληθυσμός από το χώρο διαβίωσής του. Πρόκειται λοιπόν για τέτοιου είδους έγκλημα. Με αυτό τον απότερο σκοπό και μάλιστα αν έχουμε και συγκεκριμένους χάρτες, αν δείτε πού ακριβώς υπάρχουν τα περισσότερα θύματα, εκεί υπάρχουν περισσότε, υπάρχει περισσότερος ε, ε κασίτερος ή χρυσός. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σαφές ως κίνητρο. Αυτό που είναι όμως ατυχές είναι ότι κυρίως η γυναίκα είναι ο στόχος τέτοιου είδους ε, εγκλημάτων γιατί είναι και ο πυλώνας ε, της οικογένειας, είναι ο πυλώνας της κοινωνίας και όταν καταστρέφεται αυτός ο πυλώνας είναι πολύ πιο εύκολο να ε, εκδιωχθεί ολόκληρη η κοινότητα που αποτελεί στόχο κάθε φορά. Σε 15 χρόνια λοιπόν είδαμε σε ιατρικό επίπεδο την εξέλιξη των διαφόρων πράξεων ε, επιτόπου. Όταν άρχισε ο πόλεμος στη λαϊκή δημοκρατία του Κογκό ε, το 1996, είδαμε ότι η σύγκρουση αυτή δεν αφορούσε τόσο, τουλάχιστον είδαμε έτσι, ε, αυτή ήταν, αυτό το ιατρικό μας πόρισμα, θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί σε οποιαδήποτε ένοπλη σύραξη μετά την απόφαση του Καμπιλά να επιστρέψουν οι σύμμαχοι στις χώρες προέλευσης τους, ε, ε, μία-δύο εβδομάδες μετά υπήρξε μία αλλαγή τακτικής και η αλλαγή τακτικής χαρακτηριζόταν ε, το 1998-99 είχαμε αρχίσει, να βλέπουμε ε, ολόκληρες γυναίκες που έρχονταν με πολλές πληγές στα γεννητικά όργανα και βλέπαμε ότι ήταν οι γυναίκες οι οποίες είχαν υποστεί βασανισμό σε πολύ με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και βλέπαμε τις πληγές στα γεννητικά τους όργανα. Ε, ε, και μάλιστα βέβαια οι γυναίκες αυτές παρέμεναν ζωντανές. Μετά τις διαπραγματεύσεις ε, ε υπήρξαν ε, Υπήρξαν ομάδες ε, οι οποίες γνωρίζαμε ότι θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρξει και μία άλλη ε, ομάδα ε, του κογκολέζικου πληθυσμού, του Μάι Μάι έτσι τους αποκαλούσαμε τότε, και υπήρχαν επίσης και οι πρόσφυγες από τη Ρουάντα, οι οποίοι έχουν μια πολιτικο-στρατιωτική συμμαχία κάτι το οποίο ε, είναι τελείως διαφορετικό, θα οδηγήσει σε τελείως διαφορετική κατάσταση και θα, θα, διαπιστώσουμε τότε ότι η, ο πόλεμος είναι κοντά και κάθε φορά είναι η κοινωνία, ο πληθυσμός που ε, πλήττεται. Αυτό ε, ο πληθυσμό ε, πλήρωνε το μεγαλύτερο το τίμημα, οι άμαχοι και κυρίως οι γυναίκες. Και τότε διαπιστώνεται βέβαια ότι υπήρχαν πολλές γυναίκες που είχαν πάρα πολύ σοβαρές πληγές στο σώμα τους, ε, πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Συμφωνούμε λοιπόν με αυτές ε, τις ε, ομάδες, ε, το CNDP, το SMI και όλους όσους ανέφερα. Προσπαθούμε κάπως να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, όμως με ένα κάπως διαφορετικό τρόπο, χωρίς να γίνεται σεβαστός, να γίνεται σεβαστή νομοθεσία η μεταβατική που ίσχυε. Ε, υπήρξαν επίσης πάρα πολλές συζητήσεις ε, ε, και με την Μονίκ τότε. Ε, προσπαθήσαμε όλους να τους συμπεριλάβουμε και τους στρατιώτες της κυβέρνησης και τους αντάρτες που δεν είχαν καμία απολύτως εκπαίδευση και πρέπει να πω ότι υπήρχαν μάλιστα και παιδιά 10 ετών, παιδιά 10 ετών που μπήκαν στο Αντάρτικο 10 ετών και είχαν ε, ε, όπλα στα χέρια τους μόνο και μόνο για να μπορούν να φάνε. Ήταν ένα μέσο για να έχουν κάποια λεφτά, να έχουν κάποια τρόφιμα, να έχουν ό,τι θέλουν και βέβαια και γυναίκες. Πρόκειται λοιπόν για, μια, για, μια, ε, για παιδιά τα οποία τα ενθαρρύνουμε στο μίσος και στη βία, όμως δεν είχαμε λάβει τότε υπόψη μας αυτή την πτυχή της ε, ψυχολογικής ε, καταστροφής που υφίστανται τα παιδιά αυτά, δεν υπήρξε ποτέ ένας, ε, μια, μια προσπάθεια αποκατάστασης των ανθρώπων αυτών, των παιδιών αυτών, ώστε να ε, ξεχάσουν τα τραύματά τους και όταν θα γίνουν ενήλικοι να μπορέσουν να είναι σωστοί στρατιώτες. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, αυτό που είδαμε στο Φυζί, στον Παράκα ή σε διάφορες άλλες περιοχές, ότι δηλαδή όταν μιλάμε για FRDC, ε, δεν μιλάμε για ε, βία, αλλά δεν λέμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που προβαίνουν σε βίαιες πράξεις. Όταν βλέπετε λοιπόν τα διάφορα στάδια τα οποία σας αναφέρω εδώ, είναι νομίζω σαφές ε, και βλέπω ότι είναι πολύ σημαντική η συζήτηση. Πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση για να ξέρουμε ακριβώς ποιο κάνει τι. Σήμερα η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό δεν γνωρίζουμε καλά τον ακριβή αριθμό των γυναικών που έχουν υποστεί βιασμό. Είναι κάπως ε, ε αστοιχείωτα τα νούμερα που έχουμε ε, στην, ε, στη διάθεσή μας δεν μπορούμε συνεπώς να ξέρουμε την εξέλιξη των εγκλημάτων, πώς γίνονται τα εγκλήματα αυτά. Όταν λοιπόν ε, ε, στρατεύουμε νέους στρατιώτες, τους βάζουμε σε μια ομάδα και σε μια κοινωνία χωρίς καθόλου να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τα τραύματά τους και να τα αφήσουν πίσω τους και χωρίς να λάβουμε υπόψη βέβαια ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ποτέ μια εκπαίδευση σεβασμού των γυναικών και σεβασμού της κοινότητας στην οποία ανήκουν. Και ένα τελευταίο φαινόμενο ε, για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω είναι ότι βλέπουμε επίσης όλα τα παιδιά τα οποία είδαν τους ε, γονείς τους να σκοτώνουν και να βιάζουν, που είδαν ότι οι γονείς τους ε, δεν έτυχαν σεβασμού και τότε αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι θα συμβεί στην κοινωνία του Κονγκό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει φτάσει επιτέλους η χρονική στιγμή να δοθεί μια ιδιαίτερη σημασία σε όλους αυτούς, ε, ε, τους, ε, σε όλα αυτά τα παιδιά που είδαν τις μητέρες τους να βιάζονται, που είδαν τους γονείς τους να υποφέρουν και με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να σέβονται και εκείνα τις ε, μητέρες των υπολείπων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχουν, υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από βιασμό και τα παιδιά αυτά δεν έχουν καμία ένταξη στην κοινωνία. Ούτε ε, πολλές φορές τα έχουν αποδεχθεί οι μητέρες τους. Είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθεί κανείς την εγκυμοσύνη όταν είναι αποτέλεσμα βιασμού και χρειάζεται μια ψυχολογική υποστήριξη ώστε να υπάρξει μια σχέση ανάμεσα στο παιδί που προέκυψε από βιασμό και στη μητέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συχνά υπάρχει ένα ποσοστό μητέρων που είναι εντελώς αρνητικές στην αποδοχή του παιδιού και μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία όταν η γυναίκα θέλει να ξαναρχίσει τη ζωή της υπάρχει μια αντίδραση την οποία έχουμε παρατηρήσει. Οι γυναίκες αυτές λένε κύριε Μουκουέγγε ε, δικό σας παιδί είναι, εγώ δεν πρόκειται να ασχοληθώ άλλο, θέλω να ξαναρχίσω τη ζωή μου και δεν θέλω να ξαναρχίσω τη ζωή μου με ένα παιδί που είναι προϊόν βιασμού. Ε, και τότε ε, η οι τότε ας πούμε πολλοί γονεί θα πούνε ε, ε αυτός ο συγκεκριμένο άνθρωπος βίασε την κόρη μας ε, και εν πάση περιπτώσει γίνεται ένας ολόκληρος φαύλο κύκλος με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο παιδί να ε, είναι ένας, ένα, ένας έκπτωτος της κοινωνίας. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια στρατηγική ώστε τα παιδιά αυτά να μπορούν να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Και θα σταματήσω εδώ. Νομίζω ότι έχω περάσει τα 15 ε, λεπτά που μου δώσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Σβένσον. Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ευχαριστήσω τους επίτιμους, επίσημους ομιλητές μας για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσαν σήμερα, όπως επίσης και για την αφοσίωση και τη δουλειά που προσφέρεται ε, για να την αντιμετωπιστεί αυτή η φοβερή σεξουαλική βία στο Κονγκό. Εκ μέρου τη Επιτροπή Δημοκρατών των Γυναικών και Ισότητα των Φίλων του Κοινοβουλίου, είναι μεγάλη μου χαρά και είναι ε, ε, ε, χαρά όλων των συναδέλφων του Κοινοβουλίου που μας δίνεται η ευκαιρία να συνεργαστούμε με σας για το θέμα αυτό και που μας δίνεται ευκαιρία σήμερα να ανταλλάξουμε απόψεις. Δύο λόγια θα πω μόνο, διότι γνωρίζω ότι πολλοί συνάδελφοι, μέλη του Κοινοβουλίου θέλουν να πάρουν εδώ το λόγο. Οπότε το μόνο που θα πω είναι ότι η αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας που στηρίζεται το φύλλο αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Αυτή η επιπλέον βία στις σειράξεις αποτελεί ε, έγκλημα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί έγκλημα πολέμου. Ένα άλλο θέμα που θέλω να θέσω εδώ είναι για να, αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις ειρηνευτικές διαδικασίες υπέρ της ε, υπέρ του ψηφίσματος του ΟΗΕ 1325. Είναι σημαντικό να γίνει αυτή η δουλειά για να σταματήσει αυτή η σεξουαλική βία. Χρειαζόμαστε μια στενότερη, ισχυρότερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και με τον ΟΗΕ για να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, να γίνουν βήματα για να σταματήσει αυτή η βία η οποία αυξάνεται στις ε, συνθήκες των σειράξεων. Πρέπει να συνεργαστούμε για να σταματήσει αυτή η φοβερή κατάσταση. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε θα δώσουμε το λόγο στα μέλη, στους βουλευτές. Πήρα το λόγο για να, πάρω το, το, να μιλήσω για δύο λεπτά. Έχουμε δύο λεπτά ανά μέλος για να μην καθυστερούμε. Μπορούμε πολλά πράγματα να πούμε με δύο λόγια. Ε, ε, δόκτωρ Μουκβέντε, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Είχα πάει το 2010 στο Μουγκαβού, είχατε την ευγένεια να με υποδεχτείτε και να μου δείξετε τις εγκαταστάσεις στις οποίες εργάζετε. Επίσης, ε, μετά από αυτό, είχαμε έρθει σε επαφή, αλλά θα ήθελα να σας πω. Κάνετε μεγάλη προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί η η σεξουαλική βία κατά των γυναικών, αλλά μεγάλο, ένα πολύ μικρό μέρο από αυτήν φτάνει στι γυναίκε στην Κινσάσα και εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι απογοητευτήκαμε πάρα πολύ γιατί ουσιαστικά τίποτα, τίποτα δεν υπόθηκε στην, για τον πολλαπλασιασμό τη σεξουαλική βία. Έθεσα το θέμα αυτό στο Γιαουντέ στην περιφερειακή συνάντηση στι 28 και 29 Απριλίου που έγιναν πολύ επικοδομητικέ συζητήσει για την σεξουαλική βία η δημοκρατία του Κονγκό, ε, συζητήσεις που μεταφέρθηκαν και στο τελικό ανακοινωθέν. Έχω ακόμα ένα λεπτό, θα σας τις αναφέρω. Προσθέσαμε στο ανακοινωθέν ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου αγανάκτησαν απέναντι στην, ε, στον πολλαπλασιασμό των σεξουαλικών εγκλημάτων και στο κίνδυνο να γίνουν αυτά καθημερινή υπόθεση. Ε, το θεωρούν απαράδεκτο και πρέπει να ε, διατυπωθεί μια ξεκάθαρη πολιτική θέληση. Θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι να κυρώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή τις σχετικές ε, δια, ε, διακηρύξεις, τις σχετικές συμφωνίες και θα πρέπει να υπάρξουν ε, χώροι για τα, για τη φιλοξενία των θυμάτων σε όλες τις εμπλεκόμενες περιοχές. Λοιπόν, τώρα ολοκλήρωσα και δίνω το λόγο στην κυρία Κουρμέη. Ζήτα. Ζήτα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω Μαρκό ότι ε, αισθάνεσαι πολύ άνετα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε συνεργαστεί σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Θεωρώ ότι τα θέματα της σεξουαλικής βίας είναι η αειδιαστικότερη επίθεση ε, ε, είναι μία από τις χειρότερες επιθέσεις κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όπως όλοι γνωρίζουμε. Δύο ε, ερωτήματα έχω ως πρακτική γυναίκα. Πρώτον τεχνικής φύσεως. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχαμε την ευκαιρία να έρθει εδώ ο πρέσβης ε, του ΟΗΕ για θέματα ή ε, πρέσβης του ΟΗΕ για θέματα γυναικών. Θέλω να μου πείτε πώς συνεργάζεστε, ποια είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ σας στο σύστημα του ΟΗΕ. Και δεύτερον, γνωρίζω ότι το βασικό μας θέμα σήμερα είναι το Κονγκό και με μεγάλη χαρά άκουσα την προσωπική ε, παρέμβαση του Δ. Μουγκέμπε. Είναι πολύ σοβαρό να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ε, και βεβαίως πριν από λίγε εβδομάδε ε, διάβασα πολύ ανησυχητικά νέα για τη Λιβύη. Ο εκπρόσωπο του ΟΗΕ είπε σε μια διάσκεψη του Συμβουλίου ασφαλεία ότι οι δυνάμει του Καντάφη παίρνουν διάκρα και ε, κάνουν σεξουαλικά εγκλήματα. Ξέρω ότι αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ξέρω όμως ότι ε, αν αποδειχθεί ότι ισχύει αυτό αποτελεί έγκλημα πολέμου. Πώ μπορούμε να το παληθεύσουμε. Έχει τέτοιες πληροφορίες ε, έχουν φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσει αυτή η πρακτική. Λοιπόν, θα ε, ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις. Μην ξεχνάτε το μέγιστο των δύο λεπτών. Έκλεισε ο κατάλογος γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Ο κύριος Γκέρνς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ε, χαιρετήσω τις προσωπικότητες που έχουν έρθει εδώ και που χειρίζονται ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ κυρία ε, Μάλστρομ που ήρθατε. Ε, Βάλστρομ που ήρθατε. Ε, σας είχα γνωρίσει όταν ήσασταν επίτροπος. Ευχαριστώ κυρία Σβένσον, αλλά θέλω να πω δύο λόγια στον κύριο Μουγκέμπε ήρθατε εδώ και ε, σας απονεμήθηκε ένα βραβείο. Σας ζητήθηκε λοιπόν να πείτε δύο λόγια για το έργο της ζωής σας. Και δύο πράγματα θα αναφέρω ότι δεν μπορέσατε ε, να τα ακούσετε, που δεν μπορέσατε να ακούσετε γιατί ο Evans Έσλερ είπε στο Κονγκό που υφίστανται φρικαλαίους βιασμού δεκάδες χιλιάδες γυναίκες κάθε χρόνο, ο κύριος Μουγκάβε ε, φροντίζει τα τσακισμένα σώματα και τις ψυχές τους. Και επίσης ε, ε, το έργο αυτό είναι εξαιρετικό. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το εύρος και την ανάγκη του και υπάρχει και μια άλλη διάσταση στο έργο σας που θα πρέπει να την επισημάνουμε, ο τρόπος με τον οποίο μιλάτε για την υπόθεση αυτή. Διότι ο βιασμός ε, ε, γίνεται με διαφορετικούς τρόπους, ε, υπάρχουν ενδοεθνοτικές διαφορές που δεν ενδιαφέρουν τη διεθνή κοινότητα, που καμιά φορά δεν εμπίπτουν στο διεθνές δίκαιο και αυτές οι γυναίκες έχουν έναν συνήγορο ο οποίος ε, ακούγεται στον, ε, στον, εξω, στον κόσμο έξω από τη χώρα και θέλω να παραθέσω κάτι άλλο εδώ, κάτι που λέγεται στην Αφρική όσο δεν θα υπάρχουν ιστορικοί για τα λιοντάρια, η ιστορία των, την ιστορία των λιονταριών θα την γράφουν οι κυνηγοί. Λοιπόν, έχουμε βάλει τους κυνηγού να γράφουν την ιστορία των γυναικών αυτών που έχουν υποστεί τόσα πολλά σε αυτές τις φρικαλές συγκρούσεις που γίνονται. Ε, σας, ευχαριστούμε εκ σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων όσοι είχαν τη χαρά να παρακολουθήσουν την πορεία σας, το προνόμιο να παρακολουθήσουν την πορεία σας και πραγματικά ελπίζουμε ότι από τη θέση αυτή θα μπορέσει να περιοριστεί αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ο Φάρμα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Βάλστρομ και τον κύριο Μουκουβέβερ. Δύο ερωτήματα κυρίω για την κυρία Βάλστρομ. Τι γίνεται με την εντολή σα στο μέλλον πρώτα απ' όλα. Από ό,τι ξέρουμε περιορισμένοι στο χρόνο, αλλά από ό,τι ξέρω θέλετε να εξασφαλίσετε μία παράταση της εντολής σας να γίνει και μόνιμη στο χρόνο. Υπάρχει κάποιο τρόπο να σας βοηθήσουμε για κάτι τέτοιο. Αναφέρατε τώρα επίσης την ε, νομοθεσία για τα ορυκτά που προέρχονται από χώρες συγκρούσεων από ό,τι καταλαβαίνω υποστηρίζετε το να δεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθεσία αντίστοιχη αυτή των ΗΠΑ. Αλλά περιμένετε να υπάρξει μια πρωτοβουλία της Κομισιόν ή των κρατών μελών ή θέλετε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρουμε την πρωτοβουλία. Και επίσης μετά από αυτή τη, την ε, συνάντηση είμαι ο οικοδεσπότης του, της παρουσίασης του έργου Resolution και θα υπάρχουν οι εθελοντές οι οποίοι υποστήριξαν αυτή την πρωτοβουλία στην διπλανή αίθουσα, την Α3G3, είσαστε καλόδεκτοι εκεί. Κυρία Νεδέτσοβα, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Wallstrom και τον κύριο Μουκβέμπε για όλα τα στοιχεία που μας έδωσαν. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μουκβέμπ για το γεγονός ότι έχει παρουσιάσει το πλαίσιο των εγκλημάτων αυτών και την σημασία τους γιατί φαίνεται ότι η σεξουαλική βία έχει γίνει πραγματικό όπλο πολέμου. Και πρέπει να υπογραμμίσουμε αυτόν το σημαντικό παράγοντα. Επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τη βία. Όταν αντιμετωπίσουμε τη βία να δούμε και τις πηγές του προβλήματος, τη θέση των γυναικών, τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται η γυναίκα. Ξέρουμε τα ταμπού της σιωπής τα οποία καλύπτουν αυτό το θέμα. Τι κάνει λοιπόν το σχολείο ώστε τα παιδιά σε μια νεαρή ηλικία μαθαίνουν ότι υπάρχει ισότητα ανώ και γυναικών. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να υπάρξει συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και ιδίως και της δικαστικής εξουσίας. Τι γίνεται στο δικαστικό σύστημα ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες οι οποίες καταθέτουν να μπορούν να υπάρχουν πραγματικά παραδείγματα αν υπήρξαν κάποιοι οποίοι τιμωρήθηκαν για τέτοιου είδους εγκλήματα. Κυρία Βόλσον, για, τα για τα θύματα. Ξέρουμε το πιο δύσκολο είναι να κάνουμε τις γυναίκες αυτές να μιλήσουν. Πώς εξασφαλίζεται να υπάρχουν δομές υποδοχής με άτομα καταρτισμένα για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα και επίσης για την πρόληψη. Αν ο ΟΗΕ προβλέπει να έχει προγράμματα πιο στοχευμένα που να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα οποία άκουσα σήμερα, ιδίως για τη δραματική αυτή κατάθεση του δόκτωρα Μουγκέβε, που νομίζω ότι είναι πράγματι ένα παράδειγμα για το πώς μπορούμε με πιο καλή εστίαση και περισσότερο σε βάθος να δώσουμε έμφαση σε αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει με μεγάλη σοβαρότητα η ε, η Ευρώπη. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει και συμβολικό χαρακτήρα μέσα στην οικογένεια, έχει κοινωνικό χαρακτήρα, έχει και οικονομικό χαρακτήρα. Πρέπει να έχουμε λοιπόν περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή μας. Το πρώτο ερώτημα για μένα είναι να αντιμετωπίσουμε και την κατάσταση των παιδιών. Θα ήθελα να ξέρω αν κύριε Μουκβέγγε έχετε κάποια σχέδια και προγράμματα που φέρνουν σε πέρας μήκυο στη χώρα σας και τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο υπό την έποψη της συνεργασίας για την ανάπτυξη από την πλευρά της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεύτερον, αν θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα ελέγχου των συνόρων. Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν άτομα τα οποία έρχονται από άλλες χώρες όπως η Ρουάντα και μέσα στη γενική σύγχυση. είναι ολόκληρα χωριά τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί και έχει φύγει ο πληθυσμό από εκεί λόγω αυτού του φαινόμενου. Και επίση, ποιο είναι ο νομικός ορισμός που ισχύει στην, ε, στο Κονγκό για τη σεξουαλική βία κατά γυναικών, παιδιών, ακόμα και ανδρών. Και ξέρω ότι υπάρχουν 130 περιπτώσεις που ήρθαν ενώπιον των δικαστηρίων. Θα ήθελα να ξέρω τι έγινε ε, στις περιπτώσεις αυτές και αν υπάρχει νομοθεσία που αποτελεί, που θεωρεί ότι αυτό το αδίκημα έχει επιβαρυντικό χαρακτήρα και πώς συνδέεται με τα εγκλήματα πολέμου. Και σας υπενθυμίζω και την έρευνα της Κάρλα Ντεορπόντι για τα ζητήματα αυτά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει συνεργασία με την Κομισιόν για όλα αυτά τα θέματα. Με ενδιαφέρει η ανιχνευσιμότητα και μια καλύτερη ικανότητα ε, η Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέτει γυναίκες σε θέσεις διαπραγματεύσεων. Έχετε ξεπεράσει κατά παρασάγκα στον χρόνο ομιλίες σας και αποστερείτε άλλα μέλη της Επιτροπής από την χρήση του λόγου. Κύριε Σβένσον. Σας ευχαριστώ και με εσύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω και σας κυρία Βάλστρομ και σας δόκτωρ Μουκουβέγε Είναι κάτι το απίστευτο αυτό το οποίο ακούσαμε, αλλά το έχουμε ξανακούσει φυσικά και στο παρελθόν. Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα για σας, δόκτωρ. Τα παιδιά τα οποία έχουν αναγκαστεί να γίνουν παιδιά στρατιώτες, φυσικά έχουν ψυχικά τραύματα και έχουν σημαδευτεί από αυτή την εμπειρία για όλη τη ζωή τους. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουν αυτά τα παιδιά να νιώσουν κάποια συμφιλίωση με τον εαυτό τους και με την κοινωνία γύρω τους. Και κάτι ακόμα. Είμαι πεπισμένος ότι θα βρούμε κορίτσια και κορίτσια από όλη την ε, Αφρική μετά από αυτά τα φαινόμενα και στη Λιβύη και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει εμείς να καλωσορίσουμε όλα αυτά τα άτομα και να μην κλείσουμε τα σύνορά μας και απλώς να συζητάμε αυτό το θέμα για το τι γίνεται στο Κονγκό και κάποιες άλλες χώρες στην Αφρική. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάισνερ. Ja, Σας ευχαριστώ και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομη γιατί έχουν λεχθεί τα περισσότερα. Δεν είναι πρώτη φορά φυσικά φορά που βλέπουμε αυτά τα αποτρόπαια γεγονότα. Ένα συγκεκριμένο ερώτημα για την κυρία Βάλστρομ. Είπατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΗΕ για τα θέματα αυτά. Πώ φαντάζεστε αυτή τη συνεργασία σε πρακτικό επίπεδο, πώ θα μπορέσει να γίνει κάτι για να βελτιώσουμε τα πράγματα και για τον κύριο Μουκβέγγερ. Υπάρχει κατά την άποψή μα επαρκή ανθρωπιστική βοήθεια. Χρειαζόμαστε περισσότερου ιατρού, περισσότερη ψυχολογική υποστήριξη για τι κακοποιημένε γυναίκε και τα παιδιά ή έχετε αρκετά άτομα και δεύτερον, κατά την άποψή σας, τι θα έπρεπε να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει την κατάσταση στη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τόνσκης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να πω ότι γνώριζα τον δόκτορα Μιχφέγκε, τον ήξερα ως μεγάλο ανθρωπιστή και ε, πολύ σημαντική προσωπικότητα. Πρέπει να πω ότι τρέφω τον υψηλότερο σεβασμό για όλα όσα κάνετε. Και εγώ ως πρώην ε, καθηγητής πανεπιστημίου θα ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με τα πολιτικά μέσα και τις δυνατότητες που, μπορούμε να, με τις δυνατότητες που έχουμε να κάνουμε κάτι κατά αυτού του καταστροφικού φαινομένου στον κόσμο. Γνωρίζουμε ότι μερικές φορές ε, υπάρχει μία... Ε, το, το, γεγονός ότι υπάρχει βία σημαίνει ότι δεν είμαστε αρκετά επιτυχείς σε όλες τις προσπάθειές μας. Δηλαδή, είναι μερικές φορές δύσκολο να καταλάβουμε γιατί υπάρχει βία και συνεπώς δεν μπορούμε να είμαστε επιτυχείς σε όλα θέλουμε να κάνουμε. Πώς... Ε, ε, θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε στα εγκλήματα πολέμου ε, την, ε, τον, τον βιασμό και τη δολοφονία των γυναικών. Μήπως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στα προγράμματα των πανεπιστημίων, να, λαμβάνεται να λαμβάνετε δηλαδή υπόψη το πόσο φρικτά είναι αυτά τα εγκλήματα που γίνονται κατά των γυναικών σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Μπάουερ. Ε, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την εκτίμηση ε, ε, που τρέφω για την ε, ανταλλαγή αυτή απόψεων με την κυρία Βάλστρομ και τον κύριο Μουκουέγγε. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ευθύνη της διεθνούς κοινότητας. Γιατί μπορούμε εμείς ε, να ε, εκφράσουμε την άποψή μας. Ε, έχει κάποιο νόημα αυτό, αλλά νομίζω ότι η φωνή μας δεν εισακούεται στο Κονγκό και σε άλλα μέρη του κόσμου. Όταν, ας πούμε, γκρίνουμε κάποιο ψήφισμα. Η δουλειά του κυρίου Μουκουέγκε δείχνει και αυτά που μας είπε δείχνουν ότι ο βιασμός δεν είναι απλώς μία πράξη, σε τόσο μαζική κλίμακα ε, ε, γιατί έχουμε πληροφορίες για το πόσο μαζικό φαινόμενο είναι αυτό το πράγμα, αυτό που γίνεται στο Κονγκό, η σεξουαλική βία. Μιλάμε για εκατομμύρια περιστατικά και είναι κάτι που πραγματικά καταστρέφει τον ιστό της κοινωνίας. Επομένως, έχει μακροχρόνιες συνέπειες για ολόκληρη την κοινωνία με ιδιαίτερο στιγματισμό και βέβαια με όλες τις συνέπειες που έχει αυτός ο στιγματισμός. Οπότε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, εσείς κυρία Βάλστρομ στο, στο ε, στον ΟΗΕ και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό εξοχώτης, ε, ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, δεν ξέρω αν θέλει να πάρει το λόγο ε, για μια σύντομη παρέμβαση. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μπορείτε παρακαλώ να καθίσετε. Σας παρακαλώ καθίστε. Είμαι η πρόεδρος αυτής της συνεδρίας σας και σας ζητώ να καθίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ, κυριέ μου. Κυριέ μου, σας παρακαλώ, καθίστε, ε, βιντεοσκοπήστε αν θέλετε με την ησυχία σας, αλλά θα αφήσετε τον ε, πρέσβη να απαντήσει. Και αν δεν σας αρέσει να φύγετε από την αίθουσα. Σας δίνω το λόγο, κύριε πρέσβη. Παρακαλώ σεβαστείτε τους κανόνες ε, της ε, Επιτροπής μας. Ε, μπορείτε να βιντεοσκοπήσετε όποιον θέλετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα καλέσω την ασφάλεια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να αποχωρήσετε. Σας παρακαλώ πολύ Παρακαλώ Παρακαλώ να αποχωρήσετε. Μα τι είναι αυτή η κατάσταση. Πέρα τη συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι, πέρα τη συνεδρίαση. Παρακαλώ πολύ, καλό την ασφάλεια. La séance est Πέρα στη συνεδρίαση, παρακαλώ. Πέρα στη συνεδρίαση, κυρίε και κύριοι. La Επαναλαμβάνω, πέρα στη συνεδρίαση. Περιμένω την ασφάλεια εντωμεταξύ διακόπτουμε τη συνεδρίαση. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι απαράδεκτο. Τρία λεπτά διακοπή της συνεδρίασης, κυρίες και κύριοι.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 deux minutes à la Commission et cinq. Can you, do, can you reply in 5 minutes, do you think? Messieurs, dames, nous allons pouvoir reprendre place, s'il vous plaît. Να ξαναρχίσουμε παρακαλώ τη συνεδρίαση. Merci de prendre place et de... Καθίστε παρακαλώ και σας ευχαριστώ που κάνετε λιγότερο θόρυβο. Λυπάμαι για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και ανεύθυνη συμπεριφορά. Συγγνώμη εξοχότατε. Συγγνώμη εξοχότατε που δεν σας αφήσαμε να λάβετε το λόγο. Ελπίζω εξοχότατε να μην ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί δεν φαίνει τίποτα το θετικό. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται στη χώρα σας και προσπαθούμε όλοι να βάλουμε το πετραδάκι μας για να περατωθεί αυτή η εφιαλτική κατάσταση. Καταλαβαίνω τις αντιδράσεις ορισμένων, αλλά πρέπει κάποιοι κανόνες να γίνονται σεβαστοί είτε στη Δημοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό, είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας δίνω αμέσω το λόγο εξοχότατε, εάν θέλετε. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, να χαιρετήσω το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το επιδεινούμενο δράμα του πληθυσμού του Κονγκό. Όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν, δεν είναι κομμάτι του πολιτισμού μας. Δεν τα κάνουμε για να σκηθούμε στο εθνικό μας σπορ. Όλοι ως Αφρικανοί θέλουμε να είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε τη γυναίκα μας, τη φίλη μας, τη μητέρα μας ε, και τη συνάδελφό μας. Άρα αυτό που συμβαίνει είναι ό,τι χειρότερο, η χειρότερη κατεσχήνη για έναν άνδρα και πραγματικά αυτό που συμβαίνει πλήττει όλο τον πληθυσμό της χώρας. Προσπαθούμε να το να το δούμε χρονικά. Ο γιατρός μίλησε για 12-15 χρόνια. Η μέθοδος που εφαρμόζεται είναι ξενόφερτη και τα διάφορα ψηφίσματα από την εποχή του 1234 του ΟΗΕ μέχρι και το ψήφισμα που αφορά την εσωτερική κατάσταση στο Κονγκό για τον περιορισμό του δράματος διαπιστώνουμε ότι όλο και περισσότερο ε, έχει γίνει κάτι που δεν μπορούμε να το ανεχθούμε. Έχουν ληφθεί μέτρα και απαντώ σε μία βουλευτή η οποία ε, αναφέρθηκε σε δικαστικά μέτρα. Δεν ε, τίθεται τέτοιο θέμα Όσον αφορά την κατάπαυση των εχθροπραξιών και του διακανονισμού των γκρίζων ζωνών. Μην ξεχνάτε ότι το 1994 στο Κονγκό έφτασαν 2 εκατομμύρια ε, πρόσφυγες σε δύο εβδομάδες και ο πόλεμος διήρκεσε 10 χρόνια με τις φοβερές αυτές συνέπειες που πέσαν δυστυχώς οι γυναίκες. Άρα η λύση πρέπει να είναι συνολική, ολιστική. Αν μιλάμε για ε, τα δικαστήρια πρέπει να μιλάμε και για την ψυχολογία, την ψυχολογική υποστήριξη, για τα παιδιά που είναι στρατιώτες και που ενηλικιώθηκαν, για τις γυναίκες που έχουν χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους και όλα αυτά, κυρία Πρόεδρε, για να πούμε αυτά, να απαντήσουμε σε αυτά τα οποία λέτε. Ήρθασαν στην Κινσάσα, ε, ασχοληθήκαμε εκεί ε, με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλοί παριστάμενοι εδώ δεν ήταν εκεί. Είμαστε οι πρώτοι που έχουμε συμπεριλάβει στην νομοθεσία μας το βήμα, τον βιασμό, τον βιασμό, έτσι απλά και μόνο τον βιασμό ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί και η έννοια της ισότητας ε, διευρύνεται, οι γυναίκες παίρνουν θέση, ε, υποφέρουν. Όπως είπε και μια άλλη κυρία ε, ή όπως είπε και κάποιος άλλος, την ιστορία των λιονταριών θα τη γράφουν οι κυνηγοί όσο δεν υπάρχουν πραγματικοί ιστορικοί. Υπό την αιγίδα λοιπόν του αρχηγού του κράτους στο Κονγκό αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ολιστικά, με συνολικό τρόπο. Γιατί η γυναίκα έχει περιθωριοποιηθεί και έχει γίνει δύο φορές θύμα. Πράγμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό που κάνει ο δόκτωρ Μουγκουέγκε εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια. Χρειάζεται όμως πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η, όλο και λιγότερα εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει υποστεί τις συνέπειες. Όλο και περισσότερο η λύση ή οι λύσεις που μπορεί να είναι και συντονισμένες και αυτό σας ενδιαφέρει από το διαπιστώνω, μας οδηγούν προς τη λύση αυτού του σοβαρού προβλήματος. Ίσως θα πρέπει να συγχωρήσουμε κάποιες υπερβολές. Είμαστε σε παραμονές εκλογών στο Κονγκό και υπάρχει ε, υπάρχουν κάποιες ε, ακραίες θέσεις. Αλλά τα θύματα είναι αυτά που υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Κύριε Πρόεδρε, ε, σας ευχαριστώ που συμπεριλάβατε ε, το θέμα αυτό στη συζήτηση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε με ηρεμία να συγκρίνουμε την κατάσταση, τα νούμερα. Χτες ε, ε, ε, ακούστηκαν έπαιρνοι για αυτά που κάνει ο δόκτωρ Μουγκέβε. Σήμερα ζητώ συγγνώμη για αυτά που διαδραματίστηκαν εδώ και τα οποία είναι απαράδεκτα. Κλείνοντας κυρία Πρόεδρε θέλω να σας πω ότι είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό σε βάθος. Εγώ ξεκίνησα το δημόσιο βίο μου ως υπερασπιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είμαι εξαιρετικά ευαίσθητο στο θέμα αυτό. Θέλουμε να προωθηθεί σε επίπεδο Προεδρίας Δημοκρατίας η παρακολούθηση γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο νομικό, μόνο δικαστικό, μόνο κοινωνικό. Είναι συνολικό Μπορείτε λοιπόν να προτείνετε ίσως και στο ψήφισμα ένα τέτοιο μέτρο. Θα σας ήμασταν ευγνώμονες. Γιατί αυτή, αυτό το έγκλημα πραγματικά πλήττει την καρδιά της κοινωνίας μας και μας ταπεινώνει όλους. Σας ευχαριστώ όλους και τώρα θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν, τον κύριο Ντίκενς, για ένα λεπτό δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο ήθελα να πω από τη δική μου πλευρά είναι φυσικά να συγχαρώ τον δόκτωρα Μουκουέγγε για το βραβείο που φέρει το όνομα του Βασιλέως Μποντουέν και το οποίο το αξίζει τόσο πολύ και που δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Η Κομισιόν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο θέμα αυτό Δεν το λέω τώρα αυτό σαν πρόφαση ή σαν δικαιολογία, αλλά έχουμε ήδη προσπαθήσει να παρέμβουμε στον τομέα της δικαιοσύνης, στον τομέα της υγείας και σκεφτόμαστε να κάνουμε και άλλα. Έχουμε μεγάλη ευαισθησία για την ανάγκη να ξεπεράσουμε το στενό πλαίσιο των προσπαθειών μας για την υποστήριξη προς τη Δημοκρατία του Κονγκό για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό και προβλέπουμε τη δυνητική ενίσχυση της υποστήριξής μας προς τη δικαιοσύνη και τους άλλους φορείς. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος. Δίνω το λόγο στον ε, δόκτωρα Μουκ Βεγγέλ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη για αυτό που έγινε. Είναι λυπηρό να προσπαθεί κανείς να αντιμετωπίσει τη βία με τη βία, το να είναι κανείς μισαλόδοξος είναι, κάνει πολύ δύσκολο το να υπάρξει συμφιλίωση. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξει μια τέτοια αντιμετώπιση δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Ζητώ συγγνώμη για όλους τους κοινοβουλευτικούς. Δεν νομίζω ότι δώσαμε ένα καλό υπόδειγμα για το τι γίνεται στο Κονγκό. Υπάρχουν υπεύθυνοι άνθρωποι μεταξύ μας. Τούτου τώρα θα ήθελα να σχολιάσω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φάρμ. Πώς θα μπορούσαν αυτά τα εγκλήματα να γίνουν πιο γνωστά. Αυτό είναι κομμάτι της εργασίας μας, γιατί πιστεύω σε τελική ανάλυση ότι όταν οι συμπεριφορές αυτές έναντι των γυναικών μόνο όταν γίνουν αντιληπτές ότι η, αντιληπτό ότι αυτό εμποδίζει μια φυσιολογική σχέση με τις γυναίκες όταν υπάρχει μια τέτοια άσκηση βίας. βίας. Υπάρχουν πολιτιστικά πλαίσια, υπάρχει το εθνικό πλαίσιο το οποίο όμως δεν αρκεί για να σταματήσει αυτά τα φαινόμενα. Τα άρθρα 12, 13 και 14 του συντάγματός μας τονίζουν την ισότητα δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών στο Κονγκό. Αυτό είναι κομμάτι του συντάγματος. Αλλά όπως είπε και ο εξοχότατο κύριο Πρέσβης, έχουμε πολύ καλή νομοθεσία. Το θέμα όμως είναι η εφαρμογή τους, που είναι αυτή τη στιγμή προβληματική. Για να εφαρμοστεί η νομοθεσία βέβαια, θα πρέπει να ξεκινήσει να <clears throat> γίνεται συνειδητοποίηση πολύ νωρίς στην παιδεία, ώστε τα νεαρά αγόρια να γνωρίζουν πώς πρέπει να φέρονται στις γυναίκες. <clears throat> Νομίζω ότι έχουμε τα εργαλεία για την παρέμβασή μας στα θέματα αυτά και μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε αυτά τα εργαλεία όπως το ψήφισμα 1325. Το ψήφισμα αυτό έχει ηλικία 10 ετών. Σε πολλές χώρες όμως δεν υπήρξε ούτε καν η έναρξη της εφαρμογής αυτού του ψηφίσματος. Έχουμε λοιπόν πολύ καλή νομοθεσία, αλλά το απαραίτητο είναι να υπάρξει η σωστή συνειδητοποίηση των πληθυσμών, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και στη χώρα μου, εγώ θα ήθελα να ε, προτείνω και να υποστηρίξω να γίνεται αυτό από την πιο τρυφερή ηλικία. Η κυρία Νεντελτσέβα μίλησε για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα βέβαια, αλλά σε νομικό επίπεδο είναι κάτι το οποίο έχει καταγραφεί και καθιερωθεί. Απλώς θα πρέπει η δικαιοσύνη να απονέμεται και εκείνοι οι δυσκολίες που έχουμε. Εγώ μίλησα για την πρόληψη. Νομίζω ότι μετά από αυτά τα οποία σας είπα για, το, για τη χρονική εξέλιξη και επίσης και τα ιατρικά στοιχεία και το πώς δουν ορισμένε ομάδες του πληθυσμού. Όταν έχετε μέσα στο δάσος παραγωγός χάρη ένοπλες ομάδες από το εξωτερικό, όταν ε, βρίσκονται αντιμέτωπες αυτές οι ομάδες με γυναίκες, τις φέρνουν στο δάσος και τις κάνουν σεξουαλικούς σκλάβους. Πρόσφατα απελευθερώθηκαν 80 γυναίκες που είχαν περάσει δύο χρόνια στο δάσος σε αυτή την κατάσταση. Οι μέθοδοι λοιπόν μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με την περίπτωση. Αλλά <clears throat> είναι απαραίτητο να μπορούμε να έχουμε και ένα προληπτικό τρόπο δράσης για όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Και δεν υπάρχει επαρκής πρόληψη για τα παιδιά επίσης. Δεν πρέπει να Φαντάζεστε ότι ένα παιδί που έχει δει να κακοποιείται η μητέρα του μπορεί να σεβαστεί μια άλλη γυναίκα. Τι γίνεται λοιπόν για τα παιδιά. Νομίζω ότι μέχρι στιγμή έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Αυτοί οι οποίοι βιάζουν αυτή τη στιγμή είναι παιδιά, στρατιώτες, οι οποίοι είναι οι αντάρτες αυτή τη στιγμή και έχουν κρατήσει αυτή τη βία συμπεριφορά. και όταν έγινε η αποστράτευση ουσιαστικά των ε, ενόπλων ομάδων, κανείς δεν έλαβε υπόψη την κατάσταση αυτών των παιδιών που είχαν σκοτώσει και είχαν βιάσει σαν παιδιά κατά τη διάρκεια του πολέμου. Να απαντήσω λοιπόν το ερώτημα του αν υπάρχει επαρκής κάλυψη σε ιατρικό και σε ψυχολογικό επίπεδο, αν γίνονται όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν. Νομίζω ότι ήδη αυτά τα οποία γίνονται σε ανθρωπιστικό επίπεδο είναι αξιέπαινα γιατί το κατεπήγον είναι να σωθούν γυναίκες οι οποίες κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους, έχουν σημαντικά προβλήματα υγείας. Πάντα οι επενδύσεις που υπάρχουν θα πρέπει να αυξηθούν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και έχουμε και επίσης τα προβλήματα με γυναίκες οι οποίες βιάζονται από φορείς του AIDS και εκεί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε σύντομο χρονικό ορίζοντα τα φάρμακα κατά των ρετροϊών για να εμποδίσουμε το να μεταδοθεί η ασθένεια. Πρέπει πάντως να υπάρξει μια σύνδεση μεταξύ της ανθρωπιστικής αρρωγής που λειτουργεί πολύ καλά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ανάπτυξη και αρχίζουμε να βλέπουμε πολύ καλά ότι μια γυναίκα η οποία έχει βιαστεί, η κατάστασή της είναι πολύ σοβαρή. Αναρωτιέται κανείς πώς το άτομο αυτό μπορεί να βγει από το φαύλο κύκλο που βρίσκεται. Όταν όμως το άτομο αυτό μπορεί να είναι μέσα σε μια κοινότητα και η κοινότητα να τη βοηθήσει και δεν είναι αφημένη στην τύχη της, εκεί είναι το πραγματικό πρόβλημα, γιατί η ανθρωπιστική παρέμβαση μπορεί να σώσει μια ζωή, αλλά δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι το άτομο αυτό θα μπορέσει να ξαναβρει την αξιοπρέπειά του και τη θέση του σε μια κοινότητα όταν ζει συνέχεια με εφιάλτες. Πώς θα μπορέσει να έχει δίπλα της άτομα τα οποία θα ξαναδείξουν στο άτομο αυτό ότι έχει κάποια αξία, ότι τις έχουν προσπαθήσει να τις πάρουν τα πάντα αλλά εξακολουθεί να έχει αξία σαν άτομο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσα προβλήματα, να έχουμε λοιπόν αρκετούς ψυχολόγους οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα θύματα αυτών των βιασμών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από αυτή την άποψη χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη βοήθεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας βοηθήσει για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το συνόλο των θεμάτων που ακολουθούν την αντιμετώπιση των άμεσων και επιγουσών καταστάσεων. Και αυτό θα ήθελα λοιπόν να σας τονίσω ότι χρειάζεται μια πλήρης παρακολούθηση και περίθαψη των θυμάτων. Έχουμε μήκυο στη χώρα μας, έχουμε φορείς των Ηνωμένων Εθνών, έχουμε πολλούς φορείς που δρούν επί το το μεγάλο πρόβλημα όμως που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι το πώς θα μπορέσουν να συντονιστούν οι ενέργειες όλων αυτών των ομάδων και των οργανώσεων, να ξέρουμε ποιος κάνει τι ποιος παίρνει τη βοήθεια από ποιον και να ξέρουμε ότι αυτά τα οποία παίρνουν οι φορείς αυτοί φτάνουν πραγματικά στους αποδέκτες. Πιστεύω ότι μια παρακολούθηση και μια εποπτεία για το τι έρχεται στο Κονγκό ως βοήθεια και ε, πώς χρησιμοποιείται, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο επίπεδο θα μπορούσε να γίνει αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στην κυρία Βάλστρομ Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, δυστυχώ ε, ό,τι συμβαίνει στον πόλεμο γίνεται μερικέ φορέ τρόπο ζωή στη συνέχεια και αυτή είναι η εμπειρία μα από πολλέ ενόπλε σειράξει. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα τι ερωτήσει που μετέθησαν για τον ε, συντονισμό με την ε, UN Women. Ναι, προσπαθούμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ και υπάρχει επίσης και μια πλατφόρμα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής ε, βίας κατά των γυναικών και είναι, είναι μια πλατφόρμα στην οποία συμμετέχω και εγώ. Για τη Λιβύη, ναι, πράγματι... Ε, δεν έχουμε δεδομένα που να έχουν επαληθηθεί από τον ΟΗΕ για την ώρα. Αλλά αν περιμένουμε όλα τα αριθμητικά στοιχεία, όλα τα δεδομένα να επιβεβαιωθούν, θα είναι πάντοτε πάρα πολύ αργά για να δράσουμε. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη και στους ε, οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και στους ε, οργανισμούς του ΟΗΕ για τα στοιχεία ε, που θα μας διαθέσουν. Επίσης προσπαθούμε να αυξήσουμε την παρουσία μας επί τούτου, επιτόπου συγγνώμη, από πλευράς ε, ε, οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να εξασφαλίσουμε ότι και τίθενται τα ερωτήματα αλλά και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προλάβουμε τέτοιου είδους πράξεις ή να τις αντιμετωπίσουμε. και νομίζω ότι ε, έχουν ε, γίνει και οι σχετικές κατηγορίες ε, κατά του Καντάφη σε, και το λέω αυτό σε σχέση με αυτά που είπατε στην παρέμβασή σας. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα πρέπει να αποδείξουμε για να παραμείνω, για να συνεχίσει η εντολή στον ΟΗΕ πρέπει να, αποδείξουμε την προστιθέμενη αξία μας, πρέπει να συνεχίσουμε ενδεχομένως στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ε, αλλά ε, θα είμαστε υπόλογοι απευθείας ε, στον Γενικό Γραμματέα θα ήμουν πραγματικά πολύ ευγνώμων αν θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πιέσει προκειμένου να εξακολουθήσει να ε, υφίσταται αυτή η προσπάθεια και θα ήθελα να ενθαρρύνω ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε οποιοδήποτε επίπεδο μπορεί ε, να αναλάβει πρωτοβουλίες και για να μπορέσει να συνεχιστεί αυτό που ξεκίνησε στις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ο συνολικός στόχος είναι βεβαίως ε, να προλάβουμε τέτοιου είδους ε, διεθνή εγκλήματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που λείπει από απόψε ως διεθνούς νομοθετικού πλαισίου, ρυθμιστικού πλαισίου στις διάφορες χώρες. Το πρόβλημα δεν είναι οι νόμοι. Ε, έχουμε φιλόδοξες νομοθεσίες ε, και στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα, κατά πόσο υπάρχει θέληση και η δυνατότητα εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής, επιβολής της νομοθεσίας αυτής. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Επίσης θα ήθελα να πω ότι σήμερα βάσει του διεθνούς δικαίου η σεξουαλική βία είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ε, βασανιστήριο ή γενοκτονία. Ούτως ή άλλως δηλαδή η σχετική νομοθεσία υφίσταται διεθνώς. Νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών μέσω ενός σημείου εστίασης ε, να εξασφαλίσουμε ότι είμαστε αρκετά καλά συντονισμένη, ότι έχει ενσωματωθεί το θέμα αυτό στις πολιτικές μας και ότι σε όλες τις διαπραγματεύσεις ε, εκπροσωπούνται παρκώς οι γυναίκες. Και επίσης ε, ότι η σεξουαλική βία θα αναφέρεται ως συγκεκριμένο πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να συντονίσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο τη δουλειά μας στο μέλλον και αυτό έχει να κάνει και με την αλλαγή της φύσης ε, των ε, ενόπλων σειράξεων. Ε, οι γυναίκες πλήττονται πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Το ότι οι γυναίκες, πούμε, μπορεί να βρίσκονται στο πεδίο του πολέμου και να είναι θύματα Ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήθελα να πω. Τελικά πήρα τόσο χρόνο όσο και ο κύριος μου Κουέγγε. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Αυτή η όλο αναστάτωση συνεδρίαση ήταν τελικά επικοδομητική. Θα ήθελα να ε, σας ε, ε, διαβεβαιώσω κύριε Μουκουέγγε για τη διαθεσιμότητα τη δική μου και όλων των συναδέλφων μου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εκ μέρους των γυναικών για όλα όσα κάνετε. La séance reprend à 15 15h. Πέρα στη συνεδρίαση, ε, η απογευματινή συνεδρία στις 3 η ώρα. Στην ίδια αίθουσα.